Eh, Καλημέρα σας. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω και τους προσκεκλημένους μας. Έχουμε ήδη ένα τέταρτο καθυστέρηση. Με πάση περιπτώσει ας το χαρακτηρίσουμε ακαδημαϊκό τέταρτο. Βέβαια πρέπει να έχουμε κατά νου το ρολόι γιατί νομίζω ότι θέλουμε να τελειώσουμε όλοι στην ώρα μας και φαντάζομαι ότι και θέλουμε όλοι όσοι το επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Η σημερινή ημέρα θεωρώ ότι είναι σημαντική. Η Επιτροπή Ελέγχου προπολογισμών. το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δαπανίσει αρκετό χρόνο για να ασχολείται με τη σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στους ε, διάφορους οργανισμούς ε, και τα εξωτερικά γραφεία. Έχουμε λοιπόν την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, ε, το οποίο ήλεγξε τέσσερα γραφεία ή οργανισμούς. Η κυρία Σάντερ θα μας ενημερώσει από αυτού. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να φάω όλο από το χρόνο και δίνω το λόγο στην κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να πούμε ότι ο στόχος του σεμιναρίου είναι οι συνάδελφοι βουλευτέ και πρώτη-πρώτη εγώ να εξετάσουμε τι γίνεται στα πλαίσια της ε, απαλλαγής για την Επιτροπή και για τις περιφερειακές υπηρεσίες. Να έχουμε επομένως την κατάλληλη ενημέρωση, τόσο ώστε να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε για κάτι το οποίο όλο ένα και περισσότερο ε, είναι πιο διφορούμενο, επίμαχο, αλλά ταυτόχρονα είναι και δύσκολο και λεπτό, μια από οι βουλευτές όλοι πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε τα μέσα, τις λύσεις, ούτως ώστε να μπορούμε να διακρινόμαστε από διαφάνεια αντί του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα να μην ε, υπολοιπόμεθα σε αποτελεσματικότητα. Θα θυμάστε ότι έχουμε περιπτώσεις χτυπητές ε, συγκρούσεων συμφερόντων. Πολύ σημαντικό αυτό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οικοδόμησης. Τα θεσμικά όργανα πρέπει να αποφασίζουν, έχουν κάποιες αρμοδιότητες, αλλά ταυτόχρονα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχει κάποιο έλεγχο, κάποιο αντίβαρο σε αυτέ τι εξουσίε και αρμοδιότητε. Και πάνω από όλα διαφάνεια. Οπότε και ο κόσμο εκεί εστιάζει την προσοχή του. Τα έχουμε πει και με τον Επιτροπό Μπάνγκεμαν τότε. Και θυμάστε τι έγινε με την Ισπανική εταιρεία Τελεφώνικα. γιατί όλα τα θεσμικά όργανα προσπαθούσαν από τότε να καταβάλουν ό,τι προσπάθεια γίνεται και να συμβάλλουν στη ζήμωση που γίνεται στον κόσμο. Έχουμε επίσης και τον ε, Επίτροπο Ντάλη, ε, γιατί εκτός από αυτή την Επιτροπή ασχολούμαστε και με την τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους στην Επιτροπή των ε, Μεταφορών. Οπότε και με τον Επιτροπό Κάλλας τότε υπήρχε ε, αυτή η μεγάλη πολεμική σε σχέση με το πώς επηρέαζε τα πράγματα ε, κάποια μεγάλη εταιρεία. Τα είδαμε λοιπόν και στον τύπο των διαφόρων χωρών, οπότε και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, ε, την σύγκρουση των συμφερόντων, ούτως ώστε να δούμε πώς θα ε, υπάρχει αντίβαρο στα συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα, σε σχέση επίσης και με τα επιμέρους πρόσωπα, και έτσι να μπορούμε να έχουμε κάποιους ελέγχους και για λογαριασμό των Ευρωπαίων και από πλευράς ε, ημών των βουλευτών. Και έτσι να έρονται αυτές οι συγκρούσεις. Γι' αυτό και έχουμε κάποιους κώδικες διοντολογίας που έχουν θεσπιστεί από τα θεσμικά όργανα. Οπότε είπαμε και στον ιδιωτικό τομέα έχουμε τέτοιε σύγκρουση συμφερόντων, οπότε και εδώ συντρέχει ο κώδικας διοντολογία που έχει θεσπίσει η Επιτροπή. Έχουμε επίση και διοργανική συμφωνία και γι' αυτό το λόγο και θεσπίστηκε αυτό το μητρό κώδικας, όπως θέλετε πέστε το, για διαφάνεια για τα ευρύτερα συμφέροντα της βιομηχανίας των επιχειρηματιών, των συνδικάτων, των φορέων των ε, οικολόγων, γενικά κάθε κλάδο. Και γι' αυτό και θεωρώ ότι το σημερινό μας σεμινάριο έρχεται στη σωστή στιγμή. Τη στιγμή που θέλουμε να γίνει κάποια αναθεώρηση αυτού του μητρώου, του πρωτοκόλλου των ε, συμφερόντων. Και ακριβώ μέσα από τη ζήμωση και τη συζήτηση μπορούμε να εξαγάγουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Πέρσι δε, στα πλαίσια της ε, απαλλαγής για τις περιφερειακές υπηρεσίες και την Επιτροπή, ξεκαθαρίστηκε το τι γίνεται για κάποιες ε, υπηρεσίες. Τι γίνεται για κάποιους ε, οργανισμούς που βρίσκονται σε λεπτή θέση, γιατί έχουν εντολή που αφορά το δημόσιο συμφέρον. Από την Επιτροπή δηλαδή ή το Κοινοβούλιο για να λάβουν κάποιες αποφάσεις εκτελεστικού χαρακτήρα. Και διαπιστώθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν σημεία και περιπτώσεις όπου θα μπορούσε να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Και επομένως αυτό που θέλουμε να κάνουμε και εγώ προσωπικά είναι να δούμε πώς θα θωρακίσουμε αυτές τις ε, υπηρεσίες από αυτό το κίνδυνο και πώς θα έχουμε την προστασία που τους αυτών των υπηρεσιών από την έκθεσή τους στα συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα. Έχουμε επομένω όλε αυτέ τι υπηρεσίε που δουλεύουν παράλληλα με την Επιτροπή και έχουμε επομένω και ένα σωρό άλλε δράσει όπου ε, πρέπει να βοηθούν εμπειρογνώμονε για βιοτεχνολογία, για ε, ασφάλεια νέα κυκλοφορία, χημεία, υγεία, φαρμακοβιομηχανία και για όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι ειδικοί, κάποιοι εμπειρογνώμονε. Και εκεί επομένω μπορεί να υπάρχει κίνδυνο σύγκρουση συμφερόντων. Ακριβώς και σε αυτό το, το, το επίπεδο της μεγάλης εξειδίκευσης υπάρχει αυτός ο κίνδυνος όσον αφορά την βιομηχανία, όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, οπότε και χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Χρειάζεται να υπάρχει δήλωση σε σχέση με τα συμφέροντα και από αυτούς τους εμπειρογνώμονες, αλλά επίσης και από τα διοικητικά συμβούλια, τα μέλη τους. αναδείχθηκε κατά αυτόν τον τρόπο από πέρσι το τι δυσκολίες υπάρχουν για να υπάρχει έλεγχος, να υπάρχει διαφάνεια και ότι υπάρχει ο κίνδυνος για το πώς θα καταφέρουμε, ή ο κίνδυνος μήπως και δεν καταστεί δυνατόν, να υπάρχει ο έλεγχος αυτών των συμφερόντων από πλευράς των ε, εμπειρογνωμόνων των ειδικών, των μελών των διοικητικών συμβουλίων. Θα πρέπει να δούμε το ότι πολλές φορές αυτοί οι εμπειρογνώμονες προσλαμβάνονται απευθείας στα διοικητικά συμβούλια και όχι πάντα από την ε, περιφερειακή υπηρεσία. Προτείνονται επομένω μια σειρά λύσεων για να αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος. Το δε ε, ελεγκτικό συνέδριο απαιτεί από το Κοινοβούλιο το να προβούμε σε κάποια ανάλυση. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η ανάλυση για το τι μπορεί να γίνει για αυτόν τον κίνδυνο και πού μπορούμε να ζητήσουμε τις λύσεις. Έχουμε σε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες που μπορουμε να ζητησουμε τις λυσεις εχουμε από τον ΩΣΑ και αφορούν γενικότερα την δημόσια διοίκηση. για να δούμε τι θα γίνει με το συμφέροντα των εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα. Ό,τι κάθε φορά συντρέχει, γιατί έχουμε και σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση και με τα λόμπι και τους λομπίστες, τη βιομηχανία, σε σχέση με τις δουλειές που γίνονται με το δημόσιο, με την ευρύτερη έννοια και με το κοινοβούλιο. Άρα θα πρέπει και εμείς να έχουμε σαν βάση, σαν αφετηρία αυτούς τους κανόνες του ΩΣΑ, αλλά θα πρέπει να πάμε και παραπέρα από αυτούς, γιατί έχουν τα όρια τους αυτοί οι κανόνες. Περισσότερη διαφάνεια στη σχέση μας επομένως με τον ιδιωτικό τομέα, περισσότερος έλεγχο αυτής της σύγκρουσης συμφερόντων. Θα πρέπει πριν δώσουμε το λόγο στους εμπειρογνωμονές μας, να δώσουμε έναν θετικό τόνο, λέγοντας ότι υπάρχουν μελέτες που ξεκαθαρίζουν ότι παρά το ότι ε, ο κόσμος ε, μας κατηγορεί, θεωρεί ότι εμείς είμαστε ας πούμε το, το, το ιστορία της ιστορίας, εμείς τα θεσμικά όργανα, Καταγνύουν λοιπόν αυτές οι μελέτες ότι η έκταση, ο βαθμός ανάδειξης τέτοιων συγκρούσεων συμφερόντων είναι πολύ μικρότερος εδώ στα θεσμικά όργανα παρά στους αντίστοιχους φορείς των κρατών μελών. Παρά το ότι εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε τόσο έχουμε κάποια σκάνδαλα, έχουμε 27 κράτη-μέλη, έχουμε τα υποψήφια κράτη-μέλη, κάθε τόσο κάτι συζητιέται τέτοιο. Αυτές οι μελέτες λένε ότι δεν είναι δεν είναι εδώ τα χειρότερα. Επομένω, όχι μόνο εμεί, αλλά και το Συμβούλιο προς τα μέλη του θα πρέπει να επισημαίνει την προσοχή που πρέπει να δείξουμε για τα σκάνδαλα, τα εθνικά πέραν των ευρωπαϊκών. Θα πρέπει να αναζητήσουμε τους τρόπους για να περιορίσουμε στο μέγιστο βαθμό αυτούς τους κινδύνους. Να αναζητήσουμε κάποιους, κάποιες λύσεις, πρόληψη, ε, εκ των υστέρων επανόρθωση και αυτό θα είναι και το θέμα του σημερινού μας σεμιναρίου. Η τάση είναι όταν εμφανίζεται κάποια προβληματική κατάσταση είναι να σπέβδουμε εκ των υστέρων. Αλλά θα πρέπει να έχουμε και υπόψη μας ότι μπορούμε να προλάβουμε τα συμβάντα με κάποιους κανόνες που θα θεσπίσουμε όταν αναδεικνύονται οι κίνδυνοι. Να μην έχουμε λάθη, διαφθορά και όσο πιο περίπλοκοι είναι οι κανόνες, από την άλλη μεριά είναι τόσο πιο δύσκολο να ασκείται ο έλεγχος. Άρα είναι το παράδοξο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Χρειαζόμαστε κανόνες. Χρειαζόμαστε κανόνες συνενετικούς. Αλλά θα πρέπει αυτά τα μέσα να μας βοηθούν να κάνουμε τη διάγνωση και θα πρέπει να μας βοηθούν να μπορούμε να τους εφαρμόσουμε. Και πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη τον Ευρωπαίο πολίτη, μια που φέτος έχει κηρυχθεί η χρονιά στην οποία θα εορταστεί η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Και ο στόχος μας θα είναι, το συντομότερο δυνατό, να αποκτήσει ο κόσμος μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα γιατί δεν περνάμε τώρα και τις ε, πιο καλές μέρες ε, όσον αφορά την ευρωπαϊκή οικοδόμηση μια που προσπαθούμε τώρα και εμείς να αναθεωρήσουμε πολλά και να δούμε πώς μπορούμε να ισχυροποιήσουμε την δημοκρατία και πώς μπορούμε να θωρακίσουμε το, τη δημόσια περιουσία. Γι' αυτό και πρέπει να πετύχουμε συμφωνία συνένεση στα πλαίσια της ε, συζήτησης που θα κάνουμε κατά τη διάρκεια του σημερινού σεμιναρίου. Σας ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα το πρώτο τμήμα της ε, συζήτησής μας με τους πρώτους πέντε ομιλητές. Θα συζητήσουμε γενικά πώς μπορούμε να αποφύγουμε την ε, σύγκρουση συμφερόντων. Υπάρχουν διάφορες απόψεις πάνω στο θέμα αυτό και ελπίζουμε ότι θα μάθουμε ε, πράγματα από τους πέντε ομιλητές μας. Ο πρώτος ε, ομιλητής είναι ο Γιάννος Μπέρτοκ από τον ΟΣΑ. Θα μας κάνει μια παρουσίαση σε PowerPoint και νομίζω ότι είναι σημαντικό να ακούσουμε τι έχει να μας πει διότι αναφέρονται και οι κατευθυντήρες γραμμές του ΩΣΑ. Θα σας παρακαλούσα να περιοριστείτε σε 10 λεπτά. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτιμώ ιδιαίτερα την ε, δυνατότητα αυτή να ε, ε, μιλήσω εδώ σήμερα από πλευράς του ΩΣΑ. Θα ήθελα να τονίσω αυτό που ονομάζουμε εμείς αποδείξεις. Συλλέγουμε δεδομένα και τα αναλύουμε και συμφωνώ απόλυτα με τις εισαγωγικές παρατηρήσεις. Και σε εθνικό επίπεδο ε, το θέμα των, ε, της σύγκρουσης συμφερόντων ε, δημιουργεί πρωτοσέλιδα. Είναι πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θεωρούνται σημαντικός στόχος στο θέμα αυτό, όχι μόνο το Κοινοβούλιο δηλαδή, αλλά όλα τα θεσμικά όργανα ε, παίζουν σημαντικό ρόλο κατά τον καθορισμό διεθνών προτύπων. Και στα πρότυπα υγεία, στη γεωργία κτλ. Ε, ε, θέτει πρότυπα σε ανάλογο βαθμό λοιπόν είναι και ευάλωτα τα θεσμικά όργανα, ε, ανάλογες είναι οι δαπάνες των λόμπι για τα θέματα αυτά και η λήψη αποφάσεων ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν ξεκινάει ε, στο, στην Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν από την αρχή ήδη να, να ασχοληθούμε με το θέμα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι ε, προφανής στόχος. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και το ερώτημα είναι αν υπάρχουν ε, επαρκείς μηχανισμοί ώστε να εντοπίσουν και ε, να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά. Συμφωνώ απόλυτα ότι ε, κινητήριο δύναμη είναι η δημοκρατία, η εμπιστοσύνη στα ε, θεσμικά όργανα. Αντιμετωπίζετε λοιπόν τις προσδοκίες του κοινού για διαφάνεια, σωστή συμπεριφορά, ε, σωστή ηγεσία, να είσαστε το καλό παράδειγμα και πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφέρω κάποια χαρακτηριστικά. Εσείς ε, αναφέρατε ότι το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο χρησιμοποιεί ε, τις ε, κατευθυντήρες γραμμές του ΟΣΑ. Γιατί, διότι όχι μόνο συνεργαζόμαστε με τις διάφορες χώρες εδώ και πάνω από δεκαετία, αλλά υπάρχει και γενική συνένεση σχετικά με το πώς βλέπουν τα διάφορα κράτη τα πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά δείχνουν πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον, ε, να έχουμε διαφάνεια και πιο σημαντικά να ε, αντιμετωπίσουμε ε, τα ενδεχόμενα προβλήματα, να τονίσουμε την ευθύνη του καθενός. Δεν μιλάμε μόνο για θεσμικά όργανα γενικά, το θέμα είναι πρακτικά πώς θα λειτουργήσουν τα πράγματα. Αυτή λοιπόν η πολύ πρακτική προσέγγιση Ε, καθιστούν πρακτικό εργαλείο της κατευθυντήρης γραμμές του ΩΣΑ. είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί σε συγκεκριμένε περιπτώσει η σύγκρουση συμφερόντων. Ε, θα πρέπει ο καθένα να αναγνωρίσει ότι υπάρχει αυτή η σύγκρουση συμφερόντων και γι' αυτό έχουμε εκπονήσει ένα πρακτικό ε, κουτί εργαλείων, μια εργαλειοθήκη, έχουμε ένα checklist, μια σειρά ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσει ο καθένας. Για παράδειγμα, διαφάνεια. Τι σημαίνει διαφάνεια σήμερα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, όταν κάποιος έχει λάβει ένα δώρο, είναι διατεθειμένος εσωτερικά να αναφέρει ότι το έχει λάβει, ότι ε, είναι διατεθειμένος να το εξηγήσει αυτό στους συναδέρφους του. Και πώς αντιδράει όταν ε, το θέμα αυτό καταλήξει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πώς θα εξηγήσει κανείς στους γειτόνους του ή τους συγγενείς του ε, ότι έλαβε το δώρο αυτό. Αυτή είναι η βάση για τη διαφάνεια. Είναι ένα θέμα δηλαδή που ξεπερνάει τα όρια της ε, νομοθεσίας, της νομοθετικής ρύθμισης. Στις επόμενες πέντε διαφάνειες θα ήθελα να τονίσω αυτά που λέμε τα μαθήματα. Πέντε μαθήματα έχουμε να μάθουμε. Ε, το πρώτο είναι η συνέπεια. Οι πολίτες περιμένουν συνεπή εφαρμογή των κανόνων σύγκρουσης συμφερόντων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε όλους τους τομείς. Η διασφάλιση λοιπόν αυτή το να υπάρχει ένας κεντρικός φορέας ο οποίος να σχεδιάζει τους κανόνες, να τους εφαρμόζει και να αξιολογεί ε, την, ε, τον αντίκτυπό τους, ε, αυτό είναι απαραίτητο. Βλέπετε εδώ τις χώρες του ΟΣΑ που συμβαίνει αυτό. Σε εθνικό επίπεδο λοιπόν αυτή είναι η γραμμή της βάσης. Μπορεί να βρείτε ε, περισσότερα παραδείγματα ε, στις εκτελεστικές εξουσίες και λιγότερε στις δικαστικές ή νομοθετικές, ε, αλλά πρόκειται για μια καθιερωμένη πρακτική. Δεύτερον, ποια είναι τα καλύτερα μέτρα για να το πετύχουμε αυτό. Δεν υπάρχει ένα μέτρο που να μπορεί να τα πετύχει αυτά. Συνδυασμός μέτρων μπορεί να έχει κάποιον αντίκτυπο. Και εδώ βλέπετε σε εθνικό επίπεδο ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά μέτρα. Όταν κάποιος αναλαμβάνει κάποια δημόσια θέση, τότε ξεκινάει η όλη διαδικασία και βλέπετε ότι υπάρχει εδώ ρόλος για τις τεχνολογίες επικοινωνιών ε, ε, ε, όπως ε, επίσης για τις ε, συμβουλευτικές εργασίες. Θα ήθελα να αναφέρω ότι έχουμε μία τάση, ε, το 25% των χωρών χρησιμοποιούν περισσότερους πόρους για την αξιολόγηση, για την μέτρηση δηλαδή του αντικτύπου κατά την εφαρμογή. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό αν σκεφτόμαστε τη δημιουργία ενός νέου συστήματος. Το τρίτο μάθημα που μπορούμε να μάθουμε Πάντα υπάρχουν συνέπειες. Εδώ βλέπετε τι γίνεται στο εθνικό επίπεδο. Όλες οι χώρες προβλέπουν κυρώσεις. Και βλέπετε ότι η μεγάλη πλειοψηφία ε, χρησιμοποιούν τις κυρώσεις αυτές, ιδιαίτερα όταν υπάρχει σημαντική παράβαση. Για παράδειγμα, ε, απαγόρευση ή περιορισμοί. Ε, ε, σχεδόν καμία χώρα δεν επιβάλλει κυρώσεις όταν ε, δεν υπάρχει εντοπισμός, ε, όταν δεν γίνεται κάποια αναφορά, διότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση. Αλλά βλέπετε ότι όταν υπάρχει παραβίαση των κανόνων, τότε υπάρχουν κυρώσεις και μπορεί να είναι από πολύ σημαντικές, δηλαδή απόλυση ή μπορεί να είναι λιγότερο σοβαρές οι κυρώσεις, να είναι πρόστιμα ή αλλαγή Τη μενή μετάθεση. Ε, το επόμενο, ε, οι χώρες μαθαίνουν ότι σημαντικό θέμα είναι η ακρίβεια. Το 1 πέμπτο των χωρών ελέγχουν το αποτέλεσμα των, των οικονομικών δηλώσεων, το οποίο σημαίνει ότι πολύ λίγες χώρες προσέχουν το περιεχόμενο ε, των δηλώσεων αυτών των οικονομικών. Ε, οι περισσότερες χώρες απλά επαληθεύουν την πληρότητα της ε, δήλωσης, δηλαδή αν έχουν ε, δοθεί πληροφορίες για όλα τα στοιχεία, δεν ε, ελέγχουν όμως απαραίτητα το περιεχόμενο. Και τα τρία τέταρτα των χωρών εξετάζουν αν έχει υποβληθεί η δήλωση αυτή. Θέμα τελείως γραφειοκρατικό. Το επόμενο που έχουμε να μάθουμε είναι ότι η διαφάνεια σήμερα είναι ο κανόνας. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές χώρες δεν απαιτούν μόνο αποκάλυψη των ε, ιδίων συμφερόντων, αλλά τα δημοσιεύουν και ε, όσον αφορά ε, αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις ε, του Πρωθυπουργού, των Υπουργών ε, και του Προέδρου, των βουλευτών, των γερουσιαστών και των δικαστών. Όλων αυτών των ανθρώπων δημοσιεύονται τα στοιχεία. Και Ε, θέλουμε να μάθουμε και ποιες είναι οι καλές ε, πρακτικές. Πρέπει να επικεντρωθούμε στον κίνδυνο. Πρέπει να δούμε πού βρίσκονται οι πηγή του κινδύνου. Ε, είναι νέοι κίνδυνοι ή παλιοί, οι παραδοσιακοί δηλαδή. Δεύτερον, ε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι αυτός ο τελικός στόχος. Ο στόχος ε, κινείται, ε, διότι από τη μία θέλουμε να διατηρήσουμε την δυνατότητα λήψης αποφάσεων ε, των σχετικών φορέων, να διατηρήσουμε την, τις δεξιότητες, το δυναμικό τους. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι λοιπόν πολύπλοκο το θέμα. Και τρίτον, πρέπει να κοιτάξουμε τις λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, οι πολιτικοί σύμβουλοι, οι νομοθέτες. Πρόκειται για διαφορετικές κατηγορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Και έχω κάποια αντίγραφα που έχουν να κάνουν με την ε, σύγκρουση συμφερόντων ε, ε, και διάφορα άλλα φυλάδια που περιέχουν και τα δεδομένα που σας παρουσίασα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη ομιλία. Μιλήσατε λοιπόν για ένα, μια εργαλειοθήκη για διάφορες δυνατότητες που υπάρχουν και μιλήσατε επίσης ε, και για τις ε, παροχές που προσφέρονται. Ε, πράγματι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και αυτό συνδέεται με διάφορα συμφέροντα, συγκαλυμμένα ή όχι. Πρέπει μόνο να είναι κανεί πολύ προσεκτικό. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι πληροφορίε που μα δώσατε, πολύ χρήσιμε Και πάμε στον επόμενο διευθυντή, στον κύριο Χάρντεν, Γενικό ε, Γραμματέα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Φαντάζομαι ότι εσείς ε, θα έχετε πολύ συχνά ακούσει περιπτώσεις ε, σύγκρουσης συμφερόντων και διαπλοκή. Χαίρομαι λοιπόν που ήρθατε σήμερα κοντά μα και φαντάζομαι θα μετέχετε να μα πείτε πολλά και ενδιαφέροντα. Για 10 λεπτά Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ελέγχου Προεπολογισμών τόσο διότι οργάνωσε τη σημερινή ημέρα, όσο και διότι κάλεσε τον ε, διαμεσολαβητή να εκπροσωπηθεί και αυτός ε, στη σημερινή συζήτηση. Θα ήθελα λοιπόν στην ομιλία μου να σας παρουσιάσω δύο πράγματα αλλά καταρχήν ζητώ συγγνώμη γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με τις διαφάνειες που ελπίζω να λυθεί ταχύτατα. to do my Um, θα προσπαθήσω λοιπόν να σας εξηγήσω τη δουλειά του Ομπούτσμαν ο οποίος ασχολείται με ε, προσφυγές που αφορούν στη σύγκρουση συμφερόντων. Και θα ήθελα να πω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην επεκτείνουμε αυτή την έννοια ε, να μην την επεκτείνουμε πάρα πολύ αυτή την έννοια τη σύγκρουση συμφερόντων. Τώρα, από τη δική μα δουλειά θέλω να προβάλλω τέσσερα σημεία και θέλω να σας πω ότι ο διαμεσολαβητής ασχολείται με προσφυγές ε, σχετικά με κακοδιαχείριση από πλευράς ευρωπαϊκών οργανισμών. Άρα δηλαδή ο διαμεσολαβητής δεν επιλαμβάνεται της ε, συμπεριφοράς ε, μεμονωμένων Αττίνων μεμονωμένων ατόμων. Εξετάζει το κατά πόσον ένας ε, ευρωπαϊκός οργανισμός ε, διεκπαιρέωσε σωστά μια υπόθεση. Άρα δηλαδή ο διαμεσολαβητής δεν είναι επιτροπή διοντολογίας που να κρίνει τη συμπεριφορά μεμονωμένων ατόμων. Όσον αφορά λοιπόν στο πρώτο από τα τέσσερα σημεία της ε, δουλειάς του διαμεσολαβητή είναι ότι οι οργανισμοί δεν μπορούν να απεκδίονται των ευθυνών τους απλά ζητώντας από τα άτομα να δηλώνουν ότι δεν ε, είναι εμπλεκόμενα σε σύγκρουση συμφερόντων. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ε, οι μεμονωμένοι άνθρωποι έχουν την ευθύνη να δηλώνουν πλήρως τα συμφέροντα που εκπροσωπούν. Αλλά και ο ίδιος ο οργανισμός πρέπει να δηλώνει κατά πόσον υπάρχει σύγκρουση και πώς προτίθεται να τον αντιμετωπίσει. Δεν θα πω βέβαια σε λεπτομέρειες. Ε, μπορείτε να δείτε τις ε, αναφορές που έχω και τη βιβλιογραφία Στι διαφάνειε που προβάλλονται αν θέλετε να ανατρέξετε σε κάποια ιδιαίτερη περίπτωση. Το δεύτερο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι ότι οι θεσμοί ε, πρέπει να λάβουν βήματα πριν ε, ληφθεί μια σημαντική απόφαση και αυτό για να μην προκληθεί εντύπωση ότι υπάρχει διαπλοκή συμφερόντων. Δεν αρκεί εκ των υστέρων να ισχυριστεί κανείς ότι ε, κατ' ουσίαν δεν ασκήθηκε επιρροή, δεν επηρεάστηκε η, λήψη απόφασης. Όπως πολύ σωστά είπε και η κυρία Γιάλε Σέντερ, το βασικότερο είναι η εμπιστοσύνη από πλευράς των πολιτών και γι' αυτό εφόσον μιλάμε για εμπιστοσύνη το φαίνεστε είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και αυτό βοηθάει και στο να ε, αποφύγει κανείς πραγματικά τη διαπλοκή. Το τρίτο το οποίο προκύπτει από τις περιπτώσεις με τις οποίες ασχοληθήκαμε είναι ότι κάποιος ο οποίος εργάζεται σε έναν ε, οργανισμό και ο οποίος διαπραγματεύεται με ε, μελλοντικούς εργοδότες, ίσως ήδη να βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων. Ε, οι κανόνες ε, που αφορούν αυτό το φαινόμενο που αποκαλούμε ως φαινόμενο κυλιόμενων πορτών, ό,τι και αν σημαίνει, προκαλεί δυσκολίες. Οι άνθρωποι λοιπόν έχουν πολλές φορές να αντιμετωπίσουν διάφορα συμφέροντα και καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα σε αυτά. Αυτή λοιπόν η άσκηση πράγματι πρέπει να λαμβάνει η χώρα και οι κανόνες πρέπει επίσης να έχουν κατά νου ότι η διαπλοκή προκύπτει όχι μόνο όταν κάποιος αφήνει έναν δημόσιο οργανισμό για να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ή αντίθετα, αλλά όταν δουλεύει κάποιος ήδη σε έναν δημόσιο τομέα και διαπραγματεύεται το τι θα κάνει μετά όταν φύγει. Αυτό που θέλω να πω αφορά κυρίως ε, υποθέσεις που τρέχουν και αφορούν στη σύσταση ομάδων εμπειρογνωμόνων και άμεσα εμπλεκόμενων. Ε, πράγματι είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφήνεια για το κατά πόσον τα μέλη αυτών των ομάδων ορίζονται ως ε, εκπρόσωποι και στην περίπτωση αυτή αυτό που έχει σημασία είναι τα εκπρόσωπα, τα συμφέροντα που εκπροσωπούν ή κατά πόσον ορίζονται ως εμπειρογνώμονες κατόπιν τούτου η σχέση τους με έναν συγκεκριμένο οργανισμό μπορεί πράγματι να ερμηνευτεί ως σύγκρουση συμφερόντων που πρέπει να αποφευθεί. Να πω και κάτι άλλο. Ο χειρισμός ε, της σύγκρουσης συμφερόντων είναι ένα καθοριστικό στοιχείο της ε, καλή διακυβέρνησης και της ε, δοντολογικά σωστής συμπεριφορά αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα της ε, ηθικής και της ιδεολογίας έχουν άμεση σχέση με τη διαπλοκή. Δεν πρέπει λοιπόν να ε, διευρύνουμε κατά πολύ τις έννοιες αυτές ε, για να καλύψουμε άλλες υποθέσεις που δεν είναι απαραίτητα σύγκρουση συμφερόντων. Για να είμαι λιγάκι πιο συγκεκριμένος, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω λίγα λεπτά αναφερόμενο σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Και θέλω όμως πρώτα απ' όλα ε, να, να διευκρινίσω κάτι. Η δική μας προσέγγιση στον ορισμό της σύγκρουσης συμφερόντων όπως και η προσέγγιση του ελεγκτικού συνεδρίου, η δική μας προσέγγιση ε, παραπέμπει σε μια βασική ιδέα του ΩΣΑ, που είναι ότι η σύγκρουση συμφερόντων έχει σχέση με καταστάσεις κατά τις οποίες ε, τα ιδιωτικά συμφέροντα και δημόσιοι λειτουργοί δίνουν την εντύπωση, και αυτό που ακολουθεί το βάζω μέσα σε παρένθεση γιατί είναι σημαντικό, δίνουν την εντύπωση ότι δημιουργούν σύγκρουση με την ε, σωστή άσκηση των καθηκόντων τους. Τέλος της παρένθεσης. Έτσι λοιπόν, σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να μην σημαίνει απαραίτητα ε, ίδιο συμφέρον του δημόσιου λειτουργού, αλλά μπορεί να σημαίνει ε, και κατ' επέκταση και οικογενειακά συμφέροντα, αν θέλετε, ή άλλου είδους ε, συμφέροντα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την ε, απόδοση του δημοσίου λειτουργού. Η σύγκρουση συμφερόντων, λοιπόν, αναφέρεται αναλυτικά την ε, δεύτερη αρχή που έχει για τον δημόσιο λειτουργό, που είναι η δεύτερη αρχή, η ακαιρεότητα. Δεν θέλω να σας ε, διαβάσω ε, όλα αυτά που αναφέρονται σε αυτή την αρχή, αλλά εδώ υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στη δεύτερη και στην τρίτη παράγραφο της σύγκρουσης συμφερόντων. Αυτό λοιπόν πρέπει κανείς να το εξετάσει μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο και των άλλων αρχών, κυρίως ε, της πρώτης αρχής που αφορά την αφοσίωση και η αρχή αυτή αναφέρει ότι ο δημόσιος λειτουργός θα πρέπει να έχει κατά νου ότι οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης υφίστανται για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Ένωσης και των πολιτών τους και κατόπιν τούτου οι αποφάσεις τους πρέπει να εντάσσονται μόνο σε αυτό το πλαίσιο. Πάμε τώρα στο τρίτο, στην τρίτη αρχή της αντικειμενικότητας. Ο δημόσιος λειτουργός θα πρέπει να είναι αντικειμενικός, ανοιχτός στις αποφάσεις του ε, και να προβαίνει σε συγκριτικές αξιολογήσεις, πάνω σε αυτές ε, να βασίζει τις αποφάσεις του ε, και σε άλλους παράγοντες που καθορίζονται όμως με απόλυτη σαφήνεια από τον νόμο. Το να μην χειρίζεται κανείς αυτέ τις αρχές, καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη για την ακαιρεότητα των δημοσίων λειτουργών. Αυτό όμω πάλι δεν σημαίνει ότι την έννοια τη σύγκρουση συμφερόντων πρέπει να την διευρύνουμε τόσο πολύ που να ε, καλύπτει τα πάντα. Και τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη περίπτωση που σας υποσχέθηκα ότι θα σας παρουσιάσω. Πρόσφατα λοιπόν εμείς ε, κληθήκαμε να εξετάσουμε μια προσφυγή κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με την έννοια ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι και μέλος του αποκαλούμενης ομάδας των 30. Ο προσφεύγων λοιπόν υπενήσεται ότι η τράπεζα πρόβησε κακοδιαχείριση διότι δεν ζήτησε από τον πρόεδρό της να αποχωρήσει από αυτήν την ομάδα των 30. Και υπενήσεται επίσης ότι αυτή η συμμετοχή υπονομεύει την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία που είναι καθοριστική για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και επίση υπενήσεται ο προσφεύγων ότι εδώ σαφώς και υπάρχει σύγκρουση ε, συμφερόντων. Εξετάσαμε λοιπόν αυτή την προσφυγή εντελεχώς. Ε, καταλήξαμε στο ότι δεν υπάρχει ε, κακοδιαχείριση. Αυτή η απόφαση εκδόθηκε στις αρχές αυτού του έτους. Η απόφαση του διαμεσολαβητή δεν αναφέρεται τόσο στη σύγκρουση συμφερόντων. Αναφέρει το γεγονός ότι το επενήσεται αυτό ο προσφεύγων, αλλά η δική μας ανάλυση δεν βασίζεται σε ε, σύγκρουση συμφερόντων. Γιατί? Διότι υπάρχει ένα πράγμα το οποίο καθιστά απόλυτα σαφές ο διαμεσολαβητής, ότι δηλαδή η θέση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, το να συμμετέχει ο πρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε μια ομάδα όπως αυτή είναι των 30, τότε η συμμετοχή του η δουλειά του δεν είναι με την ε, ιδιωτική του ιδιότητα. Άρα σύγκρουση ανάμεσα σε ιδιωτικά συμφέροντα και την επίσημη ιδιότητα, αυτό δεν υφίσταται, διότι η συμμετοχή απορρέει κατά κάποιον τρόπο από την επίσημη ιδιότητα, βέβαια με κάποιους περιορισμούς. Καταλήγοντας λοιπόν λέμε ότι ας μην ε, επεκτείνουμε την ε, έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων τόσο πολύ ε, έτσι ώστε να παρισφρεί αυτή η ερμηνεία ακόμα και σε άλλους τομείς όπως είναι η ακεραιότητα και η αμεροληψία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χάρντεν. Νομίζω εδώ υπάρχουν και κάποια διδάγματα τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου και πάμε τώρα στην Τίναμ Γιάκοπ η οποία είναι ενεργεία διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινη Πόρη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εσείς έχετε φέρει μία διαφάνεια, παρακαλώ. Thanks. Εγώ, θα το ξανά. Ε, αυτό το ε, έχουμε σε χαρτί, σίγουρα. Α, είναι, αυτό το έχουμε σίγουρα σε χαρτί. Ναι, αυτή είναι πάρα. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Η Τίναμ Γιάκοπ. Τίνα μου. Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Good morning. Thank you. Καλημέρα σας πρώτα πρώτα και ευχαριστούμε που καλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να σας δώσουμε τις εμπειρίες μας στα πλαίσια της διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων. Πρώτα-πρώτα, από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλω να σα πω ότι έχουμε υψηλή προτεραιότητα δώσει στο θέμα τη επαγγελματική ηθική. Και ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μπορέσουμε να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο τέτοια ε, επαγγελματική ηθική. Και πιστεύουμε ότι όπως έχει σήμερα το σύστημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τα μέσα στη της για να αντιμετωπίσει τις ε, προκλήσεις που προκύπτουν κάθε μέρα. Για να σας εξηγήσω πρώτα πρώτα έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων. Και τους εφαρμόζουμε στην Επιτροπή. Κάτι το οποίο έρχεται να ε, ταιριάξει με αυτό το οποίο είπε ο εκπρόσωπος του ΩΣΑ Ότι δηλαδή επενδύουμε σε προσπάθεια, σε ενέργεια και σε χρόνο στην συνειδητοποίηση. του θέματος και σε αυτά τα πλαίσια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη 100% να μοιραστεί την εμπειρία της με όλα τα θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Now, when I said that raising is key, I would never... Όταν σας είπα ότι θα θέλουμε να προσέξουμε τη συνειδητοποίηση, τότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την βασική αρχή τους ε, κανόνες που είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό αν κανείς δεν έχει κανόνες θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει κανείς να προστατολιστεί μέσα σε αυτόν τον λαβύρινθο ε, μιας καταστάσεως που μπορεί να ανακύψει ποτέ έχουμε συγκρούσει συμφερόντων και επί του προκειμένου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για όλα τα θεσμικά οργανωτικά και Έχουμε το καταστατικό για το προσωπικό που ισχύει για όλα τα θεσμικά όργανα και υπηρεσίες. Είναι σαφής η ρύθμιση και έτσι μπορείτε να διαπιστώσετε ότι θα πρέπει μια υπηρεσία, θα πρέπει ένας ε, υπάλληλο να ε, είναι ανεξάρτητος, ε, αντικειμενικός, πιστός, αμερόληπτος και βεβαίως αυτό καλύπτει και το ότι όλοι θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες και τις αρχές που έχουν να κάνουν με την αποφυγή συγκρούσεων συμφέροντων ή την διαχείρισή τους. Βεβαίω έχουμε και τον δημοσιονομικό κανονισμό που είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο αλλά δεν θα μας απασχολήσει σήμερα το πρωί. Οπότε αν ρίξετε μία ματιά σε αυτούς τους κανόνες που θα τους ε, δούμε χωριστά, πώς θα καταλάβετε το, ότι μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ε, περιπτώσεις κατά τις οποίες ε, μπορεί κανεί να αμφισβητηθεί για κυριότητα κάποια υπηρεσίας ή κάποιου υπαλλήλου. Όπως είπαμε, ε, οι κανόνες μας είναι πλήρες και καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα. Για να δούμε τώρα τα, τις εφαρμογής αυτών των κανόνων. Βεβαίω, όλες οι υπηρεσίες και όλα τα όργανα, ε, το καθένα φέρει την ευθύνη της εφαρμογής αυτών των κανόνων. Έτσι προβλέπεται από το σημερινό σύστημα και οπότε τώρα δύο λίγο να σας εξηγήσω πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταλήξει στην ε, εκπόνηση της θέσπιση αυτών των κανόνων. Θα θυμάστε ότι παλαιότερα, αλλά πιο συγκεκριμένα το 2008, εμφανίστηκε, δημοσιοποιήθηκε η ανακοίνωση Κάλλας που Διατύπωση την ανάγκη τον έχουμε ε, ψηλά στάνταρ, ψηλά πρότυπα επαγγελματική ηθικής. Επιτρέψτε να σα ξεκαθαρίσω ότι μιλούμε τώρα για τους κανόνε οι οποίοι ισχύουν για το υπαλλήλου, για το προσωπικό. Μιλούμε για τους επιτρόπους, τους πολιτικού, οι οποίοι αποτελούν άλλη κατηγορία και διέπονται από άλλη διοντολογία, άλλους κανόνες. Ερχόμαστε λοιπόν στους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής και αυτό το οποίο κάναμε επίση. το 2004 ήταν να λάβουμε μια απόφαση όσον αφορά τις εξωτερικέ ε, δράσεις, ε, εξωτερικά καθήκοντα ε, και αυτή η απόφαση ρυθμίζει διάφορε περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιο. υπάλληλος κατά τη διάρκεια της θητεία του ή όταν αποχώρησε από αυτή αναλαμβάνει κάποια άλλα καθήκοντα, κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, οπότε και έχουμε καθυντήριες γραμμές σε σχέση με ε, τα δώρα, σε σχέση με τη φιλοξενία που προσφέρεται στους υπαλλήλους μας. Και πέρσι δε το ε, ε, 2012 6 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε κάποιες ε, καθεντήρες γραμμές 6 το 10 του 2012 όσον αφορά την καταγγελία φαινομένων διαφθοράς. Επίσης, έχουμε ένα κώδικα διοικητικής διοντολογίας του 2000. Πάρα πολύ σημαντικό κείμενο και αφορά ε, την συμπεριφορά των ε, υπαλλήλων ευγένεια, και αποτελεσματικότητα που πρέπει να τους διακρίνει. Επίσης, έχουμε συγκροτήσει κάποιο είδους υποδομή της ηθικής αυτής και έχουμε επίσης ε, κάποιους υπαλλήλους οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι σε καθηγενική διεύθυνση ε, με το να φροντίζουν την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των κανόνων και προτύπων ηθικής συμπεριφοράς. Πάντως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι κάνει πολλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το θέμα της ε, συνειδητοποίησης, της ενημέρωσης, όσον αφορά τα σεμινάρια για τους νέους προσλαμβανομένους. Το 2012 έχουμε προβεί επίσης σε πάνω από 40 παρουσιάσεις και σεμινάρια εκπαίδευσης στις γενικές διευθύνσεις. Επίσης, υπάρχουν πολλές πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Να, ένα από τα πάρα πολύ σημαντικά σημεία στο οποία εστιάζουμε την προσοχή μας. Πέραν επομένως των κανόνων, ε, η συνειδητοποίηση, η ενημέρωση σε σχέση με την ύπαρξη αυτών των κανόνων και επομένω έτσι ε, διατυπώνουμε το γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, οι υπάλληλοι και η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τηρούν αυτούς κανόνες επίσης. Βεβαίω και χρειάζεται να υπάρχουν και κάποιοι, κάποιες κυρώσεις όπως ξέρετε έχουμε το EDOC που είναι ε, μια υπηρεσία επιφορτισμένη με τις πειθαρχικές κυρώσεις. Έχουμε την υπηρεσία κατά της απάτης, την OLAF, καθώς επίσης και την υπηρεσία IAS. Φυσικά, τα πάντα επιδεχόνται βελτίωση και αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Πάντως, όσον αφορά το πλαίσιο το οποίο ισχύει, δεν ξέρω αν θα έχουμε διαψεύσει ο συνάδελφος από ε, τον ΩΣΑ. Νομίζω όμως, λέω, ότι αυτό το πλαίσιο το οποίο έχουμε αντιστοιχεί στα όσα έχει προτείνει, συστήσει ο ΩΣΑ. Επίσης, να δούμε με λίγα λόγια γιατί είναι σημαντικό να υπάρχουν αυτοί οι κανόνες. Διότι έτσι θεσπίζεται κάποιο δίκαιο. Έτσι θεσπίζονται κάποιες υποχρεώσεις. Φορούν κάποιες γενικές υποχρεώσεις ότι δηλαδή υποχρεούνται οι υπάλληλοι να ενεργούν ε, πλήρη αμερόληψία και να έχουν μόνο το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά νου και όποτε βρεθούν σε περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων τότε έχει ο κάθε υπάλληλο την υποχρέωση αυτό να το γνωστοποιεί στην υπηρεσία και τότε η υπηρεσία να λαμβάνει τα μέτρα που πρέπει. το καταστατικό τώρα, πάει ακόμα παραπέρα. Προβλέπονται εκεί συγκεκριμένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες είναι πάρα πολύ πιθανό να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Και γι' αυτό, πέραν των γενικών έρχων έχουμε και συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι συντρέχουν. Εάν κάποιος υπάλληλος έχει αναλάβει να κάνει κάποια εξωτερική δραστηριότητα είτε πληρώνεται για αυτήν είτε όχι θα πρέπει σε μια περίπτωση να ζητήσει την άδεια προς τούτο. Επίσης οι δραστηριότητες των συζύγων θα πρέπει να δηλώνονται ούτως ώστε να λαμβάνονται τα τυχόν μέτρα που την υπηρεσία χρειάζεται Αυτό έχουμε και την ε, ατομική δήλωση σύγκρουση συμφερόντων. Δεν σα αναφέρω όλες τις υποχρεώσεις και όλες τις περιπτώσει τι οποίες ε, αναφέρει το κανονισμό. Πάντω, ο οργανισμό είναι αρκετά συγκεκριμένο. Τι ισχύει, αν αποχωρήσει από την υπηρεσία ε, κάποιο υπάλληλο και θέλει να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Θα πρέπει τότε να ενημερώσει σχετικά την υπηρεσία και αυτό είναι το άρθρο 16 του καταστατικού. Οπότε και το θεσμικό όργανο θα εξετάσει για να κρίνει εάν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων και είναι κάτι το οποίο θίγει τα συμφέροντα του θεσμικού οργάνου, οπότε και τότε πάλι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρο, το οποίο θα πρέπει να διαποτεθεί από αναλογικότητα. Εκτός μικροφώνου ο πρόεδρος. Ναι, ναι, δεν θα αργήσω, αλλά καθίστε να, να ολοκληρώσω αυτή τη, τη γενική άποψη των πραγμάτων. Έχουμε επομένως, ε, κανόνες οι οποίοι ε, απαγορεύουν το να εκμεταλλευτεί κανείς τις πληροφορίες που παίρνει από την υπηρεσία. Βλέπουμε ότι μας παίζει ο χρόνος, οπότε πάμε παρακάτω και είπαμε πρώτα πρώτα είναι πάρα πολύ σημαντικοί οι κανόνες. Δεύτερον, πάμε στο ότι οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται και σε αυτό το πλαίσιο θέλω να σας εξηγήσω σύντομα το ότι δυνάμει του άρθρου 16 από τότε που πρόκυψε αυτό το θέμα το, τον της σειρωμένης πόρτας ε, ότι προσπαθούμε συστηματικά με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες να το δούμε γιατί να δούμε το ότι οι τελικά λαμβανόμενες αποφάσεις θα πρέπει τελικά να χαρακτηρίζονται από αναλογικότητα και ισορροπία. Από τη μία μεριά των συμφερόντων του θεσμικού οργών και από την άλλη μεριά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το δικαίωμα στην εργασία. Δεν μπορεί κανείς λοιπόν φεύγοντας από την υπηρεσία να πει ε, όχι ε, ε, ας πούμε, να πούμε ε, δεν θα πρέπει κανεί να πάει να δουλέψει να, την ειδικότητά του. Θα μπορούσε κανεί να πει βέβαια ότι τον, τον πληρώνουμε για να μην δουλέψει δύο χρόνια, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι το πιο δόκιμο. Και από την άλλη μεριά βέβαια έχουμε και τα συγκεκριμένα ε, πειθαρχικά μέτρα. Θα πρέπει επομένω, είπαμε, να εφαρμόζονται οι κανόνε, αλλά δεν αρκούν. Και επί του προκειμένου πρέπει να σα πω ότι έχουμε αυτή την, την υπόθεση της συνειδητοποίησης και θα πρέπει ε, κανείς να, να, είναι το πράγμα προς μίμηση. Οπότε και για αυτό, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να έχουν τα μέτρα, να έχουν την καθοδήγηση τελικά οι υπάλληλοι, ούτως ώστε να μπορέσουν ε, υπεύθυνα να μπορούν να κινηθούν σε, σε ένα πλαίσιο το οποίο το κατανοούν Και έχουμε και το τεστ της εφημερίδας, όπως το λέμε. Δηλαδή, κάτι δεν θα πρέπει να είμαι λέω ότι στους Financial Times, εάν λοιπόν έκανε κάτι κάποιος θεωρεί ότι αυτό θα το δημοσιόταν στην εφημερίδα της επόμενη μέρα. Αυτό είναι το τεστ. Οπότε τώρα, όσον αφορά τις περιφερειακές υπηρεσίες, επίσης ε, είπαμε ότι ε, θα συζητηθούν αυτά στο, στο δεύτερο πάνελ ε, στο σεμιναριό μας, οπότε τέλος πάντων εμείς ενημερώνουμε τις υπηρεσίες. Και επίσης η πολιτική που εφαρμόζουμε είναι το να συνεργαζόμαστε στενά με τις υπηρεσίες, να κάνουμε ελέγχους, ε, και επίσης να βοηθούμε τις υπηρεσίες ε, όποτε χρειάζεται εφαρμογή κανόνων. Τόσο θα τα πούμε και τα υπόλοιπα στο δεύτερο πάνελ. Για ανθρώπους σαν και εμένα ή μάλλον για τους ανθρώπους που με γνωρίζουν ε, θα γνωρίζουν ότι ήμουν πάρα πολύ γενναιόδωρος εδώ σήμερα αλλά έχοντα ε, κατά νου και την ισορροπία ανάμεσα στα δύο φύλλα, θα ήθελα πολύ να σα έχω δώσει ε, για περισσότερη ώρα το λόγο. Ε, περνάμε στον επόμενο ομιλητή μας που αντικαθιστά την συνάδελφό του Γιάννα Μίτερμαϊερ που από ό,τι κατάλαβα ασθενεί. Η... Την κυρία ε, Γιάννα Μίτερμαϊερ ε, αντικαθιστά ο κύριος Ρόνι Πάτς. 10 λεπτά έχετε παρακαλώ. Καλημέρα. Μια σειρά ερωτήσεων μας τέθηκαν σε προετοιμασία αυτού του, ε, του σημερινού εργαστηρίου, του σημερινού σεμιναρίου. Ε, το πρώτο έχει να κάνει με ε, το, τον, την αυστηρή ή χαλαρή ρύθμιση και το άλλο ε, θέμα είναι αν περισσότεροι κανόνε ε, επιφέρουν μείωση τη σύγκρουση των συμφερόντων. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη σειρά ερωτήσεων. Βλέπουμε μια σειρά τάσεων. Η σύγκρουση συμφερόντων γίνεται αποδεκτή σε όλα τα επίπεδα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε εθνικό όπως και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η αναγνώριση αυτή υπάρχει τώρα και Εάν δείτε τι δουλειά κάνει το γραφείο της ε, Transparency International, ε, Διεθνής Διαφάνεια, ε, ασχολούμαστε όταν μιλάμε για τον κώδικα συμπεριφοράς των ευρωβουλευτών, των εμπειρογνωμόνων ή όπως ασχολείται ένα συνάδελφό μου με τους ανθρώπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ε, ε, μιλάμε για πολύ συγκεκριμένη νομοθεσία, για παράδειγμα την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Κάτι που ακούει κανείς συχνά στις συζητήσεις αυτές είναι ναι, αλλά η σωστή παρακολούθηση ε, απαιτεί νέους φορείς, νέα χρηματοδότηση, η γραφειοκρατία είναι πρόβλημα και έτσι συχνά αντιμετωπίζουμε την ίδια συζήτηση παρότι όλοι λένε ότι δεν είναι καλό πράγμα η σύγκρουση συμφερόντων και θα πρέπει να αποφεύγεται. Αυτή λοιπόν είναι η τάση που βλέπουμε να υπάρχει. Ταυτόχρονα ε, έχουν αλλάξει οι σταδιοδρομίες. Ε, οι, ε, τα, τα θεσμικά όργανα βασίζονται περισσότερο σε εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη, αναθέτουν μελέτες σε, σε άλλους. Έτσι λοιπόν ε, ο όγκος συγκρούσεων συμφερόντων αυξάνεται. Το θέμα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την σφαίρα που συνεχώς διωγγώνεται. Από την άλλη μεριά, η βλέπουμε έναν κόσμο που έχει όλο και περισσότερες δυνατότητες να είναι διαφανής, που έχει νέα μέσα ώστε να δημοσιεύει αυτά που πρέπει να δημοσιεύονται. Από την άλλη, τα θεσμικά όργανα αργούν να προσαρμοστούν στα σωστά εργαλεία διαφάνειας. Εάν δει κανείς το το ότι οι δηλώσει των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωβουλευτών ε, δημοσιεύονται ω PDF σε ένα σωρό διαφορετικέ ιστοσελίδε. Ε, ε, ή τα διάφορα θεσμικά όργανα, το καθένα έχει το δικό του σύστημα. Εγώ λοιπόν ως πολίτης, ως δημοσιογράφος, δεν είναι εύκολο να τα εξετάσω όλα αυτά. Το να γνωρίζω λοιπόν τι ακριβώς ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι δύσκολο. Νομίζω λοιπόν ότι η πρόκληση είναι να καταλάβουμε ότι υπάρχουν νέα μέσα και να χρησιμοποιήσουμε τα νέα αυτά εργαλεία ώστε ε, να καταστήσουμε δυνατή την δημοσίευση των ε, στοιχείων αυτών. Να μην χάνω χρόνο. Νομίζω ότι η συζήτηση σχετικά με την αυτορύθμιση σε σχέση με την πιο αυστορή ρύθμιση έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ότι η αυτορύθμιση λειτουργεί ε, θεωρητικά, στην πράξη όμως δεν λειτουργεί. Και το πρόβλημα είναι η παρακολούθηση. Το μεγάλο πρόβλημα δηλαδή είναι εάν έχουμε ήπιους κανόνες αυτορύθμιση και ελαφρύς μηχανισμούς παρακολούθησης, πώς μπορούν ε, αυτοί που ε, ε, δουλεύουν με αυτά να, να ισχυρίζονται ότι χρειάζεται περισσότερο προσωπικό, περισσότερους πόρους. Πώς λοιπόν μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεκτές να παρακολουθούν. Οι συνάδελφοί μας στο Ηνωμένο Βασίλειο έκαναν μια μελέτη σχετικά με τις περιστρεφόμενες πόρτες, το Revolving Doors, ε, γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο να αλλάζει κανείς σταδιοδρομία ενώ ε, το παραδοσιακό μοντέλο είναι ότι όλοι παραμένουμε στην ίδια θέση δημοσίου υπαλλήλου όλη μας τη ζωή και παρακολουθούμε ένα τον άλλον. Αυτό το παλιό μοντέλο λοιπόν μπορεί να λειτουργούσε παλιά, σήμερα όμως δεν λειτουργεί πια. Κατόπιν έχουμε το θέμα του αν οι περισσότεροι κανόνες οδηγούν σε λιγότερες παραβιάσεις παραβάσεις. Ε, το θέμα είναι ότι ακούσαμε ότι στο, στην Κομισιόν υπάρχει ε, ένα καθορισμένο πλαίσιο. Υπάρχουν οι απαραίτητοι μηχανισμοί ε, για την επιβολή των κανόνων αυτών. Δεν νομίζω ότι ισχύει απαραίτητα αυτό και όταν διαβάζω εγώ τους κανονισμούς αυτορύθμισης. Ε, βλέπω ότι υπάρχουν ε, πολύ ωραίες αρχές, αλλά ε, δεν νομίζω ότι ανταποκρίνονται στις προθέσεις. Δεν είναι αρκετά ισχυροί οι κανόνες αυτοί. Και τελικά, όταν ακούμε ότι η Κομισιόν προτείνει νέους κανονισμούς για ε, του, τις επιχειρήσεις, θεωρούν ότι όταν θεωρούν ότι χρειάζεται περισσότερη ρύθμιση αλλά δεν θέλουν να δώσουν εντύπωση ότι δημιουργούν περισσότερη γραφειοκρατία, λένε ότι πρόκειται για ευφυή ε, νομοθεσία. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερου κανόνε, χρειαζόμαστε ευφύ ε, νομοθεσία ώστε να μπορούμε να ε, φροντίζουμε να, να επιβάλλονται οι κανόνε. Και του χρόνου έχουμε ευρωβουλευτέ πολύ πρώην σύμβουλοι που εργάζονταν σε γραφεία υπουργών ή σε γραφεία επιτρόπων θα ε, αποχωρήσουν από το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, θα βρουν νέες σταδιοδρομίες και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε αν ε, θα λειτουργήσουν οι παρόντες κανονισμοί. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι χρήσιμο να γίνει αυτό και θα κλείσω εδώ. Ευχαριστώ. πολύ καλά. Αναφερθήκατε σε όλα τα συγκεκριμένα θέματα, απαντήσατε τις ερωτήσεις ε, και περνώ το λόγο στον επόμενο ομιλητή, τον Wolfgang Rau, ε, που είναι γραμματέας της Γκρέκο. Um, σας ευχαριστώ πολύ για το θερμό σας ε, καλωσόρισμα. θέλω και εγώ να μιλήσω λιγάκι για αυτό το θέμα της διαφθοράς. Το Γκρέκο είναι αρκτικό λεξο και δεν έχει σχέση με την αξιολόγηση ε, ευρωπαϊκών ε, θεσμών, όχι ακόμα τουλάχιστον, ίσως αυτό να συμβεί στο μέλλον, γιατί γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης στον οργανισμό Γκρέκο. Δεν θέλω λοιπόν να μιλήσω για, οργανικούς, για ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τη σύγκρουση συμφερόντων. Ο δικός μας ο ρόλος είναι να ελέγχουμε την συμβατότητα των κρατών μελών με έξι κανόνες κατά της διαφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης υπάρχουν και οι συστάσεις ε, του Συμβουλίου των Υπουργών για τον κώδικα συμπεριφοράς των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ε, νομικό εργαλείο πάνω στο οποίο βασίζουμε τις αξιολογήσεις μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 49 κράτη-μέλη, προφανώς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε επίσης ε, και τις Ηνωμένε Πολιτείε και τη Λευκορωσία. Εμείς είμαστε ο μόνος το μόνο μόρφωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε ως πλήρες μέλος και αυτές δέχονται τις αξιολογήσεις με τον ίδιο ακριβώ τρόπο όπως και όλα τα άλλα μέλη μας. Ε, στη δουλειά μας έχουμε δύο βασικούς πυλώνες. Ο ένας είναι η αξιολόγηση των κρατών μελών ε, σε σχέση με τα υπάρχοντα κριτήρια και ο δεύτερος πυλώνας είναι να ελέγχουμε σε ποιο βαθμό τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τις ε, συστάσεις που προκύπτουν από τη διαδικασία αξιολόγησης. Και αυτό είναι μια αρκετά σκληρή διαδικασία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 7 ή 8 μέλη και από το βορρά της Ευρώπης ε, που υφίστανται την διαδικασία της ε, μη συμβατότητας και αυτό γιατί τα μέλη αυτά δεν εφαρμόζουν συστάσεις που τους έχουν γίνει. Αυτό δεν έχει τόσο σχέση με την ε, σύγκρουση συμφερόντων όσο με την ε, πολιτική χρηματοδότηση. Θα επανέλθω αργότερα λιγάκι σε ορισμένα θέματα που έθιξα τώρα στην ε, εισαγωγή. Για να υπάρχει λοιπόν αποτελεσματική πρόληψη της διαφθοράς, εμείς τονίζουμε ότι στα κράτη-μέλη υπάρχει μία προϋπόθεση, δηλαδή να υπάρχει αντικειμενική αξιολόγηση των κινδύνων. Εμείς είναι γνωστό ότι, υπάρχει, ότι κάνουμε συστηματική ανάλυση παραγόντων κινδύνου, γιατί αυτό έλειπε στα κράτη-μέλη. Η σύγκρουση συμφερόντων ε, δεν ισούται απαραίτητα με τη διαφθορά, αλλά είναι ένα στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στη διαφθορά αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Παραδείγματο χάρη, κατά την, τον δεύτερο γύρο αξιολογήσεών μα, εμεί μεταξύ άλλων αξιολογήσαμε τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη-μέλη για να παρεμποδίσουν τη διαφθορά στη δημόσια διοίκηση. Ε, τις ρυθμίσεις δηλαδή που υπάρχουν για να εντοπιστεί σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα ε, στο δημόσιο και το ίδιο όφελος ε, του δημόσιου, δημοσίου υπαλλήλου. Υπάρχουν κάποιες ε, γενικές διατάξεις ε, που ισχύουν στα κρατημέλη και θελήσαμε να δούμε τις ε, συμβατότητες και να επαναλάβουμε την αρχή ότι είναι απαράδεκτο να βρίσκεται κανείς σε, εμπλεγμένο σε σύγκρουση συμφερόντων και παράνομα να εμπλέκεται και σε άλλες δραστηριότητες. Αλλά συμφωνούμε με την άποψη ότι αυτό δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να λυθεί μόνο σε επίπεδο μεμονωμένου υπαλλήλου. Οι θεσμοί ε, στους οποίους υπάγεται ο υπάλληλο και αυτοί προφανώς φέρουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Οι ρυθμίσεις που υπάρχουν για να διαπιστωθεί η ε, σύγκρουση συμφερόντων οι ε, δραστηριότητες είναι ότι ο υπάλληλος πρέπει να ενημερώσει ε, τον προϊστάμενο ή κάποια άλλη αρμόδια αρχή για το τι ακριβώς ε, συμβαίνει και ανάλογα με την κατάσταση ε, πρέπει να καταθέσει το πόθεν του. Όσον αφορά λοιπόν την αποτελεσματικότητα τέτοιων δηλώσεων, ο οργανισμός μας Γκρέκο έχει συστήσει αρκετές περιπτώσεις ε, να γίνονται πιο αυστηρές οι διαδικασίες για την επαλήθευση αυτών των δηλώσεων. Σε ορισμένα κράτη-μέλη, παραδείγματος χάνει στη Ρουμανία, εκεί έχει εισαχθεί ένα πολύ φιλόδοξο σύστημα δηλώσεων πόθεν αλλά στην αρχή δεν υπήρχε δυνατότητα να ε, διασταυρωθούν αυτές οι δηλώσεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, επί του θέματος αυτού με το θέμα αυτό ασχολήθηκε ένας άλλος εθνικός οργανισμός. Δεν θέλω να ε, δείξω ιδιαίτερα, να προσβάλλω ιδιαίτερα τη Ρουμανία, απλά το ανέφερα ως παράδειγμα. Επίσης αποδώσαμε ιδιαίτερη σημασία και στην μετακόμιση ε, των δημοσίων υπαλλήλων ε, στον ιδιωτικό τομέα, αυτό το περίφημο φαινόμενο ε, ανακυκλούμενων θυρών όπως το αναφέραμε προηγουμένως. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί ορισμένοι υπάλληλοι να ε, αποκαλύψουν ε, πληροφορίες στον νέο της εργοδότη, στον δυτικό φορέα και αυτό σημαίνει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Κατά τον τρίτο γύρο αξιολογήσεων εμείς κάναμε μία σειρά συστάσεων για να ενισχύσουμε αυτό το σύστημα των ε, κυλιόμενων θυρών, τη μετακίνηση δηλαδή παλιών από το δημόσιο στον δυτικό τομέα και αντίστροφα Υπάρχουν πολύ λίγες χώρες ε, στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Δανίας και της Ιδίας, παραδείγματος χάρη, που ε, είναι αρνητικές ε, στη ρύθμιση γιατί πιστεύουν ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό να γίνεται κάτι τέτοιο, δηλαδή οι δημόσιοι πάλι να μετακινούνται στον ιδιωτικό τομέα γιατί θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους. Άρα δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα επί του οποίου δεν υπάρχει ε, σύμπτωση απόψεων και όσους ελέγχους και να κάνουμε δεν θα επιτύχουμε τη συνένεση. Θα μπορούσα να σας αναφέρω και άλλα παραδείγματα, αλλά δυστυχώς αυτά δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο της ε, σημερινής μας συνάντησης. Θα αναφερθώ τώρα στη σύγκρουση συμφερόντων ε, στο πλαίσιο των δικών μας αξιολογήσεων. Εμείς έχουμε σχέση με την αποφυγή της διαφθοράς ε, όσον αφορά βουλευτές, ε, δικαστές και εισαγγελείς. Δεν είναι αυτό το αντικείμενό σας σήμερα, αλλά το θέμα των βουλευτών είναι κατά την άποψή μας καθοριστική σημασία. Και αυτό διότι έχει σχέση με την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς. Δυστυχώς λοιπόν τα πολιτικά κόμματα και οι βουλευτές ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν χαίρουν απόλυτη εμπιστοσύνη, χαίρουν περιορισμένη εμπιστοσύνη θα έλεγα. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Δηλαδή πώς θα ε, προβάλλουμε περισσότερο τη διαφάνεια σε σχέση με τους ε, βουλευτές. Αυτός λοιπόν ο γύρος αξιολόγησης είναι αρκετά καινούριο, ε, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012 και γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω ακριβώς ε, τι συμβαίνει. Δεν υπάρχουν ε, σαφή συμπεράσματα για όλα τα κράτη-μέλη. Όμως αναμφίβολα έχουμε αποκτήσει πληροφορίες για διάφορες καταστάσεις που αντιμετωπίσαμε. Η Γκρέκο, ο οργανισμός μας, ε, έχει αναφέρει διάφορες απόψεις ε, για το πώς πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί έτσι ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά τους βουλευτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, με μεγάλη ανησυχία, διαπιστώσαμε ότι οι βουλευτές ε, είχαν ίδιο συμφέρον κατά την σύνταξη των ψηφισμάτων και γι' αυτό ε, επικρίθηκαν και κατακρίθηκαν ε, κυρίως ε, η Πολωνία για το ότι δεν αποκάλυψαν τις προθέσεις τους. Η Πολωνία ήταν μία από τις πρώτες χώρες που αξιολογήσαμε. Βεβαίως παρεμφερεί συμπεράσματα είχαμε και για άλλες χώρες. Οι βουλευτές πρέπει να ανταποκρίνονται στη διαφάνεια να υπάρχει ώστε δυνατόν μεγαλύτερη ε, αποκάλυψη των προσωπικών του στοιχείων. Και αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τα δώρα αλλά και τις ε, φιλοξενίες. Και θα σας αναφέρω άλλο ένα παράδειγμα από μια πρόσφατη αξιολόγηση που κάναμε. Στην Εσθονία, στο Κοινοβούλιο, εκεί δεν είναι ήθιστο να καταγράφονται τα δώρα. Γι' αυτό λοιπόν απευθυνθήκαμε σε μια παλαιότερη, είδαμε μια παλαιότερη διάταξη που έλεγε ότι μπορούν βέβαια να καταγράφονται στο κοινοβούλιο τα δώρα. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτή τη δουλειά θα την κάνει ένας εξωτερικός φορέας ή θα την κάνει το ίδιο το κοινοβούλιο. Ε, και κατά πόσο το Κοινοβούλιο πρέπει να καταρτίζει τους κανόνες. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών πιστεύει ακράταντα ότι αυτό πρέπει να γίνεται στο ίδιο το Κοινοβούλιο για να διασφαλίζεται η ιδιοκτησία και για να καθίσατε σαφές ότι οι κανόνες αυτοί είναι ε, κοντά στην πραγματικότητα, όσο γίνεται βέβαια, και είναι πολύ σημαντικό τα ίδια τα κοινοβούλια να καθορίζουν μηχανισμούς για να ελέγχουν τη συμβατότητα με τους κανόνες. Μία άλλη σημαντική πρόκληση που έχει σχέση με τη σύγκρουση συμφερόντων και αυτό ήδη αναφέρθηκε αφορά τις ε, συμφωνίες ε, που συνάπτουν οι βουλευτές με τρίτα μέρη ε, και είναι πολύ σημαντικό διάφορα συστήματα δεοντολογίας αυτή τη στιγμή προστατεύουν τους ε, βουλευτές, αλλά θα πρέπει να βοηθούν έτσι ώστε να ε, διευκρινίζονται οι σχέσεις των βουλευτών με ομάδες ε, εκπροσώπησης, ομάδες πίεσης. Πρέπει να πω ότι για μας αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει μητρό των ομάδων πίεσης, να καταγράφονται αυτές. Ε, βέβαια μπορεί κανείς να καταλήξει και σε διαφορετική προσέγγιση, πάμε χάρη στη δική μας, σύμφωνα με την οποία μπορούμε να ζητήσουμε από τα κοινοβούλια να καθορίσουν κανόνες για τους βουλευτές για το πώς πρέπει να αντιδρούν αυτοί απέναντι σε τρίτη μέρη και ομάδες πίεση. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου παραδείγματο χάρη δεν υπήρχε καμία υποχρέωση για τους βουλευτές να αναφέρουν επαφές τους ε, με τρίτους ε, πέρα από συναντήσεις που είχαν σε επίσημες ε, συναντήσεις όπως συνέβη στην Πολωνία. Εμείς λοιπόν έχουμε απευθύνει μια συγκεκριμένη σύσταση στην Πολωνία αλλά δεν ισχύει και για άλλες χώρες. Δεν θα μιλήσω για δικαστές και εισαγγελείς, η κατάσταση εκεί είναι ε, παρεμφερής. Εμείς πιστεύουμε ότι οι κώδικες συμπεριφοράς και οι εσωτερικοί κανόνες οι οποίοι εξετάζουν την ασυμβατότητα και πολλά άλλα ε, συναφή στοιχεία ε, μειώνουν τις, τους κινδύνους ε, που συνδέονται με τη σύγκρουση συμφερόντων. Και έτσι λοιπόν προκύπτει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη όσον αφορά την ακαιρεότητα ε, κατά τη λήψη αποφάσεων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό να εξεταστεί το θέμα αυτό ε, και να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να εφαρμόζονται και σωστά οι κανόνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ε, σας ευχαριστούμε. Ε, και τώρα αν θέλετε ε, μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις. Δεν ξέρω ποιος από εσά επιθυμεί να υποβάλει ερώτηση. Παρακαλώ. Ε, τώρα εσείς κάθεστε στη θέση του ΕΛΚ. Αυτό θέλω να σας πω. Στα να που κανονικά κάθεται το ΕΛΚ. Ελπίζω αυτό να μην έχει καμία πολιτική σημασία ότι μεταπηδήσατε σε άλλο στρατόπεδο. Ε, ευχαριστώ. Μέρικέ Μερικές φορές συμφωνούν οι πράσινοι με το ΕΛΚ. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί εμπειρογνώμονες ε, και θα ήθελα να σας θέσω μια ερώτηση που ενδιαφέρει ιδιαίτερα ε, την Κομισιόν. Έχει να κάνει με τον διορισμό του Μισελ Πιτή ως Προέδρου της Επιτροπής Ηθικής. Επαναδιορίστηκε ως πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής, η οποία είναι αρμόδια για τον οδικό χάρτη, για την συμπεριφορά των ε, επιτρόπων. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων στο ότι ε, ήταν στην ε, νομική υπηρεσία της Κομισιόν, κατόπιν ε, εργάστηκε ως δικηγόρος και ήταν σύμβουλος ε, της βιομηχανίας καπνού και ιδιαίτερα της Φιλίπ Μόρις, η Μισελ Πετίτ. Κάποιος λοιπόν, συγγνώμη, ο Μισελ Πετίτ δεν ε, είναι περίεργο να προσλαμβάνεται αυτός για ε, την εκπόνηση του δοτικού χάρτη της συμπεριφορά των ε, επιτρόπων. Επίσης, από κάποιους δεν ζητείται δήλωση της των οικονομικών του συμφερόντων, παρότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στι εργασίες τη Κομισιόν. Και όταν μιλάτε για κυρώσεις, πού θα τις βρούμε αυτές. Ο Γενικός Διευθυντής της, ε, ε, Επιτροπής, ε, της Υπηρεσίας Φαρμακών, ο κύριος Λούντκρεν, πριν το κάνει αυτό, είχε δημιουργήσει μια εταιρεία συμβούλων που εργάζονταν σε διάφορα φαρμακευτικά εργαστήρια. Δεν επιβλήθηκε καμία ποινή. Το σύστημα λοιπόν που αναφέρεται δεν είναι αξιόπιστο μέχρι να αναγκαστεί κάποιο ε, να πληρώσει τι κυρώσει, ε, δεν θα τον σταματήσει τίποτα να ε, συνεχίσει να φέρεται με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να εκπονείται ένα σωρό κανόνες, αλλά δεν χρησιμεύουν και σε πολλά. Θα ακούσουμε όλες τις ερωτήσει μαζί και μετά θα απαντήσουν οι εμπειρογνώμονε. Υπάρχει κανεί άλλο που να θέλει να πάρει το λόγο πέρα από αυτού που ανέφερα. Ε, και σας παρακαλώ μην μακρηγορήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρωτού να έρθω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ε, ήμουνα σύμβουλος στην Ουαλία για πολλά χρόνια. Τέθηκε λοιπόν το θέμα της σύγκρουση των συμφερόντων. Ήταν ένα θέμα που ανέκυπτε και ήταν πάντα ένα δύσκολο θέμα να αντιμετωπίσουμε. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις. Το η μία έχει να κάνει με την δήλωση των συμφερόντων. Ένα θέμα το οποίο ε, συχνά αντιμετωπίζουμε είναι το αν οι ανώτατοι αξιωματούχοι θα πρέπει να δηλώνουν ε, αν είναι μέλη ε, οργανισμών, ιδιαίτερα μυστικών οργανισμών και το θέμα είναι αν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική ή προαιρετική η απάντηση. Το προφανές θέμα είναι οι μασόνοι, ε, κάποιοι λοιπόν ε, θεωρούν ότι το να δηλώνει κανείς ε, ότι είναι μέλος, θα πρέπει, ότι είναι μασόνος δηλαδή, θα πρέπει να είναι προαιρετικό. Και το άλλο θέμα θα πρέπει... Διότι κάποιες επιχειρήσεις Το, θέμα που, το άλλο θέμα που τίθεται είναι η ε, φιλοξενία. Θα πρέπει να δηλώνεται κάθε φορά ή ε, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο. Ευχαριστώ. σε ποιον απευθύνεται την ερώτησή σας. Οποιοςδήποτε μπορεί να απαντήσει. Πρέπει να υπάρχει μια εξισορρόπηση Κοιτάξτε, εγώ δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω ακριβώς αυτά που είπε η εκπρόσωπος της Κομισιόν. Το θέμα είναι ε, κατά πόσο να αρκούν οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί αυτή τη στιγμή για τον εντοπισμό της σύγκρουσης συμφερόντων. Να μας πείτε ναι ή όχι. Γιατί εμείς ε, το εξετάσαμε το θέμα αυτό ε, κατά την δική μας τη δουλειά για επεξεργασία νέων κανονισμών. Δεν ξέρω όμως ποια είναι η δική σας άποψη. Αυτό που με ενδιαφέρει επίση είναι τι πιστεύετε σχετικά με τις προτάσεις ε, που έχει υιοθετήσει και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων επιτέλους, ως ανά θα έλεγα, και σας ευχαριστούμε και πολύ. Όσοι έχουν λοιπόν ε, αυτή τη στιγμή οι κανόνες, αυτό που εντυπωσιάζει είναι το εξής. Οι υψηλόβαθμοι υπάλληλοι όταν αποχωρούν. Ο Πτήτας που, που είχε κάνει μια συμφωνία με τη Φίλιπ Μόρι και τώρα εργάζεται για την εταιρεία αυτή. Πρέπει κανείς ε, πράγματι να ψάξει αν όλα βαίνουν καλώς. Από τη θέση του ε, διαμεσολαβητή ε, συνεπέραν ότι εδώ δεν τίθεται μόνο θέμα σύγκρου συμφερόντων αλλά και ακαιρεότητας επί τη υπάρχουν βέβαια διάφορες απόψεις. Κατά την άποψή μου εδώ σαφώς είναι και θέμα σύγκρουση συμφερόντων. Οι ευαισθησίε ε, ποικίλουν. Ε, αλλιώ ορίζει ο ένα την ακερότητα και αλλιώ την ορίζει κάποιο άλλο. Εγώ θα προτιμούσα να υπάρχει μια πιο σαφή νομική βάση. Ερωτώ λοιπόν, πιστεύετε ότι αρκούν οι κείμενοι κανόνες. Ε, τι πιστεύετε για τις θέσεις τις οποίες υιοθέτησε, όπως είπα και η Νομική Επιτροπή, ως θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και δεύτερη ερώτηση, Μισελ Πετίτ. Μήπως θα πρέπει να το ψάξουμε λιγάκι. Αυτό είναι μια ερώτηση προς όλους. Τι πιστεύετε εσείς. Και το τρίτο σημείο αφορά στις σχέσεις με τις ομάδες πίεσης. Το ξαναείδαμε αυτό στην περίπτωση του Επιτρόπου Ντάλι. Μήπως ε, χρειαζόμαστε νέους κανόνες και αυτή είναι μια ερώτηση προς όλους. Ε, χρειαζόμαστε νέους κανόνες είναι μια ερώτηση που αφορά όλους ε, τους ομιλητές. Η κυρία Λεπάζ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη που καθυστέρησα να δεν μπόρεσα να ακούσω όλες τις εισηγήσεις, αλλά θα ήθελα να σας τονίσω τα εξή. πρωτα Πρώτα-πρώτα, το θέμα δεν είναι πόσους κανόνες έχουμε, είναι το τι κυρώσεις υπάρχουν, τι έλεγχος, τι εφαρμογή υπάρχει. Ένας κανόνας που δεν εφαρμόζεται, δεν έχει κυρώσεις, δεν υπάρχει. Μπορεί να κάνουμε λίστες ολόκληρες, καταλόγους. Εάν δεν υπάρχει έλεγχος και επιβολή κυρώσεων, δεν ωφελεί προς τίποτα. Άρα, θέλουμε αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, να σταματήσουν τα παραλαμβανόμενα σκάνδαλα τα οποία υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Να σταματήσει η λίστα των κανόνων. Για μένα αυτό είναι το βασικό. Βλέπετε ότι Όλα αυτά τα που έχουμε δει, τα, τα είπε και η Μισελ, είμαι 3,5 χρόνια ευρωβουλευτή. Όλες αυτές τις ανομαλίες. Θα το πούμε έτσι, διπλωματικά. Όλα αυτά τα οποία εδώ και τέσσερα χρόνια έχουν εμφανιστεί. Πάντοτε, πάντοτε όλα αυτά καταγγέλλονται απ' έξω από κάποιες ενώσεις προσώπων ε, ε οι ασθενείς, οι γιατροί, ε, από εμά του βουλευτέ, ποτέ, ποτέ από το εσωτερικό των υπηρεσιών. Άρα ο εσωτερικό έλεγχο δεν αποδίδει. Καλά δεν, δεν θα ακριβώ, ήθελα να λάβω τον λόγο κι άλλοι. Επομένω δεν είναι θέμα ποσότητα κανόνων και νόμων. θέμα είναι στην πραγματικότητα τι εφαρμογή γίνεται αυτών και τι κυρίως υπάρχουν. Δεν ξέρω τον κύριο Περιπτή Αλλά μιλούμε για κάτι συμβολικό, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο για τον Ευρωπαίο και την κοινή γνώμη. Πρόκειται για κάποια πράγματα που έχουν συμβολική σημασία. Είναι παράδεκτα και που αμαυρώνουν την εικόνα θεσμικού οργά. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο ε, πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλούσα τον ε, κύριο Ράου και τον εκπρόσωπο της ε, Transparency International να μου πει το εξής είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται εδώ. Ε, οι ευρωβουλευτές ε, δημιουργούν μια ένωση που ε, θέλει να προωθήσει τον τομέα ασφαλείας. Εδώ συμμετέχουν μεγάλοι όμιλοι από ένα κράτος μέλος. Δεν δημοσιεύεται ποια είναι ε, τα μέλη, ούτε πώς χρησιμοποιούνται ε, οι συνεισφορές των μελών ευρωβουλευτές που συμμετέχουν ε, στο Προεδρείο της Ένωσης ε, δεν το δηλώνουν ε, αυτό στη δήλωσή τους. Μάλιστα επιτρέπουν τους βοηθούς τους, βάζουν τους βοηθούς τους να δουλεύουν υπέρ τη Ένωσης αυτής πάνε ταξίδια στο εξωτερικό που δεν είναι σαφές ποιος πληρώνει τα ταξίδια και υπό ποια ιδιότητα εμφανίζονται εκεί. Εν μέρει εμφανίζονται ως βουλευτές και εν μέρει ως μέλη της Ένωσης αυτής. Η Ένωση αυτή, παρότι δημιουργήθηκε αποκλειστικά από ευρωβουλευτές, δεν, δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των λόμπις. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ακούσω εσείς πώς ε, εκτιμάτε μια τέτοια δομή. Ευχαριστώ πολύ. Ο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα, συγχαρητήρια προ την εισηγήτρια τη συνάδελφου Αγγέλα Σέντερ γιατί διάλεξε ένα πραγματικά δύσκολο ζήτημα, θέμα. Πάρα πολύ καλά μα τα είπαν οι εμπειρογνώμονες, οι ειδικοί. Δεν ξέρω τώρα, μήπω έχουμε λάθο μεθοδολογία. Γιατί συμφωνώ με την ανάλυση που έγινε από τη συνάδελφο για τι κυρώσει. Έχουμε ένα σωρό κανόνε. Και στην ουσία δεν ξέρω. Να ρωτήσουμε πώ είναι και η Ένωση σαν τη Γαλλία που είναι ο πρωταθλητής, ο παγκόσμιος για τους κανόνες, τα διατάγματα, τους νόμους που δεν εφαρμόζονται. Και έτσι οδηγούμεθα στην έλλειψη εμπιστοσύνη από τον Ευρωπαίο. Κυρώσεις χρειάζονται. Και επίσης χρειάζεται να υπάρχει διαχωρισμός εξουσιών. Άρα και για τη σύγκρουση συμφωνών θα πρέπει οι δημόσιες δραστηριότητε να είναι διαφορετικές από τις εμπορικές. Έχουμε μακραίων παράδοση στη Γαλλία όσον αφορά ε, το δημόσιο σε σχέση με, την, με τις απολαβές των υπαλλήλων, σε σχέση με εκείνους που θέλουν να ασχοληθούν με τέτοια δραστηριότητα, να δουλέψουν δηλαδή στο δημόσιο και να μην ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Γιατί ακριβώ είναι δυνατόν να έχουμε ε, πάρα πολλού σπουδαίου ε, μηχανικού από σπουδαία πανεπιστήμια και ε, επομένω χρειάζεται ο έλεγχο επί των βιομηχανικών ιδιωτικών δραστηριοτήτων, των διατροφικής αλυσίδας, ε, αν θα έρθει το, το Άλογα από τη Ρουμανία να βαφτιστεί βοδινό στη Γαλλία. Αυτό χρειαζόμαστε. Και εγώ επομένω νομίζω πρέπει να προβληματιστούμε για ε, μια, μια δημόσια υπηρεσία αυθεντικά ευρωπαϊκή. Να μην έχουμε τη συνδιαχείριση. Γιατί έτσι ουσιαστικά δεν υπάρχει δημόσιο. Ναι. πως ε, είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι Μα τι είναι, το, το, το, μισό Παρίσι. Άρα, να κάτσουμε και να σκεφτούμε πώς θα διαρθρώσουμε τα πράγματα και να μην τα ανακατεύουμε όλα τις δραστηριότητε και μετά να αντιμετωπίζουμε τη σύγκρουση συμφερόντων χωρίς να ασκούμε κυρώσεις. Άρα, κυρώσεις συν διαίρεση αρμοδιοτήτων. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφο Αγιά Σέντερ για αυτό το εργαστήριο το τόσο ενδιαφέρον. Επίσης, να μην, με επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι. Και η κυρία Γκρόσλερ ε, μας μίλησε για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον δηλαδή, για τα λόμπι. Ξέρετε, όταν ε, πρώτο ήρθα εδώ με πλησίασαν λομπίστες. Και να σας πω την αλήθεια, θεώρησα ότι με αναζήτησαν και πάντως έτσι, έτσι και εγώ έμαθα ήταν εμπειρία. Τέλος πάντων θα πρέπει κάπως να βοηθηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, από αυτούς που ξέρουν για να θεσπίσει κανόνες για τους ε, λομπίστες. Και ε, ξέρουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα, ξέρουμε ότι ο κάθε κλάδος προσπαθεί να διαφυλάξει τα συμφέροντά του και ξέρουμε τι γίνεται ας πούμε όσον αφορά την οδηγία για το κάπνισμα και πολλές φορές Πολλές φορές έχουμε να αντιμετωπίσουμε εκατοντάδε ε, λομπίστε εδώ στι Βρυξέλλε. Αλλά πολλέ φορέ αυτοί διαστρεβλώνουν το τοπίο. Άρα χρειάζονται κανόνε πολύ πιο σαφείς Κανόνε και για μα και για του λομπίστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι το θέμα μας είναι πολύ δύσκολο. Ιδίως όταν ε, μιλάμε σε αφηρημένο επίπεδο. Πώς θα πρέπει να δούμε το θέμα αντιστρόφως. Πώς θα προλάβουμε, πώς θα υπάρχει πρόληψη σε σχέση με την σύγκρουση φερόντων, πώς θα έχουμε επομένως ακεριότητα για τους ε, υπαλλήλους. μου λέγαμε, ε, θυμάμαι, στη Χάγη που είχα πάει με το γιο μου και θυμάμαι ήταν κάποιος που ήταν από τη ΣΕΛ και κάποιος επίσης υπάλληλο ε, αν, ανώτατος ε, από το Υπουργείο Εξωτερικών και είχαμε πάει να, να δούμε ένα ποσφαιρικό αγώνα Οπότε τι, τι πάει να πει αυτό. Ότι θα έρθει, ότι θα, θα με πιέσει, θα, θα μου ασκήσει πιέσεις λομπίστα ε, ο υπάλληλος του Υπουργείου ε, ή ο υπάλληλος ε, της ΣΕΛ. Όλα δεν είναι θέμα κανόνων, είναι θέμα ακυριότητας ατομικής. Εάν δεν υπάρχει προσωπική ηθική ακυριότητα, εάν δεν Ενεργεί, επί τη βάση της του, τότε τι να τους κάνει τους κανόνες. Μιλούμε τώρα για μία σειρά από υπηρεσίε κοινοτικέ. Και όλοι οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν εκεί δεν θα πρέπει ποτέ να εμπλέκονται ε, στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά πάλι και σε μια ιδιωτική εταιρεία δεν θα πρέπει ο υπάλληλο μια εταιρεία να πηγαίνει σε ανταγωνιστική. Πάντω είναι δύσκολο κάθε φορά να βρούμε τη διαχωριστική γραμμή, το όριο. Ε, δηλαδή πόσο θα πρέπει τελικά ε, να εξεύρουμε κάποιους ξεκαθαρούς κανόνες. Πώς θα δοθεί ο ορισμός της προσωπικής ακυρότητας, πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τους κανόνες μας ε, παντού σε όλες τις υπηρεσίες. Πώς θα γίνει αυτό. Νομίζετε ότι είναι δυνατόν μόνο με κανόνες να λυθεί το πρόβλημα. Αυτό είναι μια αυταπάτη. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλό το ότι προέκυψε μετά από την απαλλαγή πέρυσι ε, το ότι αποφασίσαμε να, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ε, θέλω να σας πω ότι και εγώ είμαι στόχος των ομάδων ποιήσης, γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι σε αυτές τις επιτροπές ε, τα μέλη του Κοινοβουλίου Προβουλευτές ε, πρέπει να έχουν ε, άποψη που να την εκφράζουν. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εγώ μετέχω σε ορισμένους οργανισμούς γιατί ε, τους συναντώ όλους ανοιχτά. τους συναντώ όταν είναι όλοι μαζί, όλοι ακούνε τι λένε οι υπόλοιποι. Όλοι έχουν την δυνατότητα αντίδραση και εγώ έχω τη δυνατότητα να αντιδράσω. Και θέλω να σα πω, αν δείτε τι τροπολογίε, χιλιάδε τροπολογιών καμιά φορά, ε, μπορείτε ε, από τις τροπολογίες να ξέρετε ποιος ευρωβουλευτής συναντήθηκε με ποιον. Εντάξει, δεν είναι και κακό αυτό απαραίτητα, γιατί αν δεν συναντά κανείς και κανένα, ε, δεν μπορεί να κάνει και τη δουλειά του. Ε, γι' αυτό πρέπει οι συναντήσεις να γίνονται ανοιχτά, με απόλυτη διαφάνεια. Εγώ αυτό κάνω και συστήνω και σε άλλους. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και θέλω να ρωτήσω το εξής Νομίζω είναι αρκετά εύκολο να εκπονεί κανείς ε, κανόνες ε, εφόσον μπορεί να εκμεταλλευτεί την εμπειρία άλλων οργανισμών ε, του και οργανισμών από άλλες υπήρους. Η ερώτησή μου αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκε ότι υπάρχουν 19 μέγιστες διασυνδέσεις. Με 19 μέγιστες διασυνδέσεις μπορεί να, να δικτυωθεί με οποιονδήποτε στον κόσμο. Ε, πώς είμαστε λοιπόν προετοιμασμένοι ε, για αυτή την εποχή, όταν δεν θα συναντάμε πια κανέναν. Απλά θα ε, γίνεται η διασύνδεση διαδικτυακά που αυτούς με τους οποίους μιλάμε μπορεί και να μην τους γνωρίζουμε, να χρησιμοποιούν και άλλο όνομα. Έτσι λοιπόν όσον αφορά στη σύγκρουση συμφερόντων, πέρα από το να ασχολούμεθα με το παρελθόν, θα πρέπει να δούμε λιγάκι και τι θα κάνουμε στο μέλλον, σε αυτή την ψηφιακή εποχή. Αν δεν τα σκεφτούμε όλα αυτά, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε και να εξετάσουμε το βασικό πρόβλημα πίσω από τη σύγκρουση των συμφερόντων, που είναι ακριβώς η έλλειψη εμπιστοσύνης. Για μένα λοιπόν η σύγκρουση συμφερόντων είναι ένα μέσο, εκείνο που έχει σημασία είναι πώς μπορεί να γεφυρωθεί, γεφυρωθεί το χάσμα ε, έλλειψη εμπιστοσύνη ανάμεσα στον πολίτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που για μένα αξίζει τον κόπο να εξάσουμε περισσότερο είναι, όπως σας είπα, τα μέσα κοινωνικής ε, δικτύωσης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ε, για τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. Ε, ακούσατε τις ερωτήσεις. Ε, δεν ξέρω, να δώσουμε πρώτο λόγο στην εισηγήτρια ή καταρχήν να απαντήσουν οι ομιλητές. Ό,τι θέλετε εσείς, λέει ο Πρόεδρος. Ίσως είναι καλύτερα να ακούσουμε καταρχήν τις απαντήσεις και μετά θα λάβετε εσείς τον λόγο. Ας ακούσουμε λοιπόν τις απαντήσεις. Αναφέρθηκε ο κύριος Πετίτ. Επίσης, το κατά πόσον λόγο ε, της ε, περίπτωσης θα πρέπει να υπάρξουν ε, οι κανόνες Επίσης ε, τέθηκαν αρκετές ερωτήσεις προς την ε, Transparency International. Έγινε και λόγος για ακυρώσεις, ε, για την ακαιρεότητα, ατομική ακαιρεότητα που είναι πολύ σημαντική για την εφαρμογή των κανόνων. Ας ξεκινήσουμε με την Κομισιόν γιατί νομίζω ότι και εσείς δεχτήκατε αρκετές επιθέσεις. Υπήρξαν αρκετά ευαίσθητα ερωτήματα που σας απευθύνθηκαν. Ξεκινάμε λοιπόν με εσά και κατόπιν θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ γιατί πραγματικά θεωρώ ότι όλα όσα είπατε και ρωτήσατε για όλα όσα συζητήσαμε αποδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι το θέμα. Το θέμα αυτό της ηθικής συμπεριφοράς για την αποφυγή της ε, σύγκρουσης συμφερόντων. Παρακαλώ επομένως να μου επιτρέψετε να σας πω. Θα ήθελα να κοιτάξω με τη σειρά που βοβλήθηκαν τις ερωτήσεις να απαντήσω σε αυτές και αν ε, ξεχάσω κάποιον παρακαλώ να μου το υπενθυμίσετε ότι σας παρέλειψα. Ξεκινώ επομένω. με την κυρία Ριβαζή για, για τον κύριο Πετήτ. Πάρα να με συγχωρήσετε. Είναι κάτι το οποίο αφορά τη λειτουργία του κώδικα διοντολογίας για τους επιτρόπους. Είναι κάτι το οποίο δεν βρίσκεται στα καθηκοντά μου, αιμοδιωτές μου, οπότε παρακαλώ να μου επιτρέψετε να μην σας απαντήσω για το συγκεκριμένο σημείο. Επίσης, κυρία Ριβαζή, είπατε ότι οι γενικοί διευθυντές θα πρέπει επίσης να προβαίνουν σε δήλωση συμφερόντων. Ναι, το κάνουν αυτό, τη δήλωση αυτή η Επίτροπη. Αλλά υπάρχει δυσαναλογία εδώ από πλευρά τη νομική βάση λόγω του ότι τα, το καταστατικό ε, από ένα σύστημα κλειστό, αυτόνομο. Τώρα, από πλευράς της ε, υπηρεσίας αυτής. Είπατε για τον κύριο Λούγκρεν. Όντως. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν κανόνες για τον διορισμό του προσωπικού τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίγνωση του θέματος. Και συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες. Και θα σας τα εξηγήσει στο δεύτερο πάνελ κάποιο συνάδελφος. Αυτά όλα για να τους βοηθήσουμε τις υπηρεσίες αυτές την υπόθεση της επαγγελματικής θήκης. Επίσης, έχω το σημειώσει τον κύριο Βουάν ε, όσον αφορά την δήλωση συμφερόντων ε, διότι θα πρέπει κανείς να δηλώνει που είναι μέλος. Αυτό να είναι υποχρεωτικό. Επίσης, ε, ελέγχθη κάτι για το κατά πόσον θα πρέπει να δηλώνεται η αποδοχή προς προτάσεις φιλοξενίας και για το κατά πόσο πρέπει να οριοθετείτε το τι μπορεί κανείς να αποδεχθεί και τι όχι. Όσον αφορά την δήλωση συμφερόντων και για το κανεί αν είναι μέλο σε κάποιο φορέα, εδώ υπάρχει κάποια διάκριση. Εάν πρόκειται για ιδιωτικό φορέα, ας πούμε κάποιο είναι μέλος κάποια θρησκευτική κοινότητας. Αυτό είναι ιδιωτική υπόθεση. Αυτό δεν θεωρείται δραστηριότητα από πλευρά του προσωπικού, από πλευρά των υπαλλήλων, το που θα πρέπει να δηλούνται. Επίση, Όσον αφορά τη δήλωση για την αποδοχή κάποιες φιλοξενίας, για το προσωπικό της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό το οποίο ε, ρυθμίζεται είναι ε, η διάκριση ότι τι γίνεται επαφορμή της ασκήσεως των καθηκόντων του υπαλλήλου. Αυτό είναι το, το κριτήριο το σημαντικό. Ας πούμε, αν κάποιος υπάλληλο ε, ορίζεται ως ε, αρχιδιαπραγματευτής για κάποια εμπορική συμφωνία, ας πούμε, με τον Καναδά. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητα, η κανδική κυβέρνηση, ας πούμε, θεωρεί κομμάτι των διαπραγματεύσεων το ότι θα πρέπει ο υπάλληλο να πάει σε κάποιο δείπνο. Να, ποια είναι η διάκριση στην οποία προβαίνουμε. Γιατί για του υπαλλήλου μα τουλάχιστον κατανοούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δηλώνεται η αξία των ε, γευμάτων που προσφέρονται. Ας πούμε κανένας δουλεύει σε ε, ε, κάποια, κάποια πρεσβεία, να το πούμε και κάτι πιο ελαφρύ, εάν επομένως τον καλέσει ο, ο πρέσβης στην πρεσβευτική κατοικία, ε, πώς θα κάτσει να υπολογίσει, να δηλώσει το πόσο ωφελήθηκε οικονομικά από αυτή την ε, πρόσκληση. Είναι πρακτικό το θέμα. Κυρία Γκρέσλε. Μας μιλήσατε για τις προτάσεις, της συζητήσεις στο Κοινοβούλιο επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε δεδομένα τι απόψει των κοινωνικών επιτροπών, οπότε θα πρέπει για άλλη μια φορά να ζητήσω την κατανόησή σα ότι πρόκειται για ένα θέμα πάγιο, ε, ανοιχτό. Οι επαφέ, οι συζητήσει αυτέ συνεχίζονται. Στον αφορά το, το καταστατικό. Οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα. Ήδη είπαμε για τον Μισελ Πετίτ και τον ε, κώδικα διοντολογίας για τους επιτρόπους. Το τρίτο θέμα το οποίο θίξατε και το έχω σημειώσει είναι τι θα κάνουμε με τους ε, λομπίστες, μήπως χρειάζονται τυχόν νέοι κανόνες. Κοιτάξτε, τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν ρίξει κανεί μια ματιά στο τι κανόνε ισχύουν για την αποφυγή στη σύγκρουση συμφερόντων, θα διαπιστώσετε ότι οι κανόνες αυτοί είναι ξεκάθαροι και εάν εφαρμοστούν ακριβώς όπως είπε η κυρία ε, Γκόσλινγκ λέγεστε ε, συμπαθάτε με ένα είπα λάθος το όνομά σας ε, μιλούμε για κάποιους επομένως για τους λομπίστες θα πρέπει με διάφορο τρόπο κανεί να συναλλάσσεται με του λομπίστε. Δεν μπορεί να μείνει στον Ευαίνινο πύργο ένα υπάλληλο. Μπορεί να του συναντήσει κάποιο ε, στο δημόσιο χώρο, να του προσκαλεί στο γραφείο του. Και φυσικά με, τα αναγκαία δέοντα μέτρα προφύλαξη. Κυρία Λεπάζου, θίξατε κάτι άλλο. Το θέμα των κυρώσεων. για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι η υπηρεσία ΕΙΝΤΟΚ είναι πάρα πολύ δραστήρια. Και πρόσφατα είχαμε ένα, ένα πρώην υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης ε, Γεωργίας που ερευνήθηκε ως ομοδοσυρωτές του από την ε, Όλαφ και τελικά καταδικάστηκε σε φυλάκιση από ένα βελγικό ποινικό δικαστήριο. Άρα να προσέξουμε να μην γενικολογούμε υπερβολικά λέγοντας ότι δεν έχουμε κυρώσεις, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Αυτό πιστεύω. Τώρα και για τα σκάνδαλα τα οποία έρχονται στο φως από εξωτερικούς παράγοντες πάλι θα πρέπει να σας πω μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω ότι η βάση να επικοινωνούμε θα είναι ότι εμπιστευόμαστε τους υπαλλήλου μας ακόμα και όταν συνταξιδοτούνται. Και κατά δεύτερο λόγο δεν έχουμε τα μέσα να ελέγξουμε τα πάντα και τους πάντες. Ξέρω ότι μιλώ στα μέρη της ε, Επιτροπής των Προπολογισμών, οπότε αν τελικά αποφασίσετε ότι μπορούμε να έχουμε περισσότερο προσωπικό, τότε θα έχουμε και περισσότερους ελέγχους. Αλλά αυτό είναι δύσκολο. Δεν ξέρω τι πιέζει ο χρόνος. Νομίζω πάντως ότι τα περισσότερα τα απήντησα. Forgive me if I pronounce your name wrongly. Και επίση πάλι συμπάθεια με επιβεβαιώσω. Νομίζω οι κύριοι Οντί και Μπαλσίδη έδειξαν σημεία τα οποία κάλυψα. I too, I just see uh, one function, uh, one point which I would still like to raise. Όμως υπάρχει κάτι ακόμα που δεν το έχουμε θίξει. Και το κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε ε, τη δημόσια υπηρεσία μας και υπαλλήλου που θα, που θα έχουμε με μια προσέγγιση κάπως αμερικανική. Γιατί είναι κάποια νοοτροπία βορειοευρωπαϊκή. Δηλαδή, ένα πλήρη διαχωρισμό ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Εμεί προσπαθούμε να βρούμε να συγκεράσουμε τι απόψει, γιατί υπάρχουν αντίθετε απόψει και να έχουμε επομένω να ακολουθήσουμε τον, την εδώ. Αν κάποιο πάρει σύνταξη και κατόπιν τα όσα έμαθε για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα, τα, τα μεταδώσει σε κάποιον τρίτο και αυτό είναι χρήσιμο. Γιατί έτσι υπάρχει κάποιο είδου ε, αλληλεπίδραση αλλά αργότερα θα το συζητήσουμε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, εναπόκειται στους άλλους ομιλητές ποιος θα ήθελε να απαντήσει. Ο κύριος Ράου, παρακαλώ. Όσον αφορά την υπόθεση που μας παρουσίασε ο κύριος Ιρμάιζερ, γενικά ε, δεν σχολιάζω αυτό που εμείς στην Κρέκο θεωρούμε με μεμονωμένες περιπτώσεις. Δεν γνωρίζω την κατάσταση, δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες αλλά θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι δεδομένου ότι η Γκρέκο εξετάζει θέματα διαφάνειας στο Κοινοβούλιο, έχει τονίσει ότι Θέλουμε όχι μόνο να αποτρέψουμε, ε, να προλάβουμε τη δημιουργία ε, συγκρούσεων συμφερόντων, ε, αλλά να προωθήσουμε και την ακεραιότητα και όπως γίνεται αντιληπτή και την πραγματική. Και δεν μιλώ εκ μέρους της Γκρέκο τώρα, αλλά όσον αφορά την υπόθεση που παρουσιάσατε, αυτή η ρύθμιση δεν ε, ενθαρρύνει το κοινό να εμπιστευτεί τους ε, ευρωβουλευτές. Είναι ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει λομπίστες ε, αλλά και τρίτους και ε, είναι και αυτό κάτι που εξετάζουμε στον τέταρτο γύρο αξιολογήσεων, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ε, πέρα από τον κύκλο των επίσημων ε, ομάδων συμφερόντων, των λόμπις, υπάρχουν και πολλοί άλλοι και στην συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει σοβαρή υποψία ότι κάποιοι τρίτοι ε, προσπαθούν να, επηρεάσουν ε, αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο κοινοβουλίου. Ε, ναι, να αναφερθώ κι εγώ σε αυτό. Ε, ένας λόγος που αναφερόμαστε σε υποχρεωτικό κατάλογο των λόμπι είναι να μπορούμε να ε, γνωρίζουμε για παράδειγμα με ποιους έχουν επαφές οι ευρωβουλευτές ε, ή ε, όταν υποβάλλουν κατά λέξη τροπολογίες άλλων. Θέλουμε να αποφύγουμε λοιπόν τις μη διαφανείς περιπτώσεις. Θέλουμε δηλαδή να είναι πιο δύσκολο να είναι κανείς αδιαφανής και θέλουμε εμείς ως κοινό να μπορούμε να ελέγχουμε Περισσότερη διαφάνεια στο πολύπλοκο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθήσει τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ελέγχουν το ένα το άλλο. Δεν είμαι ε, βέβαιος εάν κάποιος γενικός διευθυντής μπορεί να γνωρίζει εάν ο υπάλληλος που τον συμβουλεύει έχει κάποιες επαφές αλλά η διαφάνεια βοηθάει όλους στο σύστημα και τον έξω και κόσμο και τα θεσμικά όργανα. Και τελικά η συζήτηση ε, καταλήγει στο θα έχουμε περισσότερο προσωπικό ε, για, τον έλεγχο. Το ερώτημα θα μπορούσε να είναι θέλουμε περισσότερο προσωπικό ώστε ε, να αντιμετωπίσουμε τα σκάνδαλα ή για να τα αποτρέψουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ απλή απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάρντεν. Uh, firstly to θα ήθελα να απαντήσω συγκεκριμένα σε αυτό που είπε η κυρία Γκρέσλερ. Να εξηγήσω ότι είπα ότι δεν θέλουμε να διευρύνουμε υπερβολικά τον ορισμό και αυτό ε, σχετίζεται με τη συγκεκριμένη περίπτωση που ανέφερα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η υπόθεση που αναφέρατε εσείς και άλλοι, κυρία Γκρέσλερ, τον πρώην Γενικό Διευθυντή της Νομικής Υπηρεσίας ε, της Επιτροπής, τον κύριο Μισελ Πετίτ. Είναι μια υπόθεση την οποία δεν είχα κατά νου και δεν εκφράζω καμία θέση σχετικά με την περίπτωση αυτή. Από ό,τι κατάλαβα, έχει γίνει προσφυγή στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για το θέμα αυτό. Μια άλλη παρατήρηση που κάνανε διάφοροι ευρωβουλευτές έχει να κάνει με τους κανόνες και το πνεύμα στο οποίο εφαρμόζονται αυτοί. Δεν μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση στην οποία οι συγκρούσεις συμφερόντων ε, ε, είναι τόσο πολύπλοκο θέμα που να ε, χρειαζόμαστε ε, γεμάτα βιβλία, γεμάτους αναλυτικούς κανόνες. Αν το κάνουμε αυτό τότε χάνουμε το βασικό νόημα το ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να αποφεύγουν την σύγκρουση συμφερόντων και τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να φέρονται με έναν τρόπο εύκολα κατανοητό σε όλους ώστε ε, να είναι διαφανή απέναντι στο κοινό. Ένα χοντρό βιβλίο κανόνων που να μπορούν να διαβάσουν μόνο εμπειρογνώμονες δεν είναι ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Η κυρία Γιάκοπ ανέφερε ότι η Κομισιόν λαμβάνει κάποιες πρωτοβουλίες ε, σχετικά με την κατάρτιση, την ευαισθητοποίηση ε, και θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερους πόρους στο θέμα ε, της σύγκρουσης συμφερόντων και μάλιστα προς αυτή την κατεύθυνση χρειαζόμαστε κανόνες, χρειαζόμαστε καλούς κανόνες, αλλά δεν χρειάζεται να τους παλοπλασιάσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, θα σας εκπλήξω μάλλον το πιο πρόσφατο μάθημα είναι ότι η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη συνδέεται με τη συμμετοχή. Τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και τη, στην εφαρμογή πολιτικών. Αυτό συμπεριλαμβάνει όλους τους βασικούς παράγοντες, όλους τους φορείς. Αναφερθήκατε στους, λο, στους λομπίστες. 80 ή 90% των χωρών θεωρούν πολύ αρνητική η δραστηριότητα το λόμπινγκ. Και η Ευρώπη δεν αποτελεί εξαίρεση. Ωστόσο, οι λομπίστες φέρνουν πληροφορίες και μάλιστα ε, παρέχουν πληροφορίες που βοηθάνε στη σωστή λήψη αποφάσεων. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ε, ισορροπία και να λαμβάνονται υπόψη όλες ε, οι απόψεις. Η σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να είναι μια προσωπική διάσταση της λήψης μιας απόφασης και μπορεί να Υπάρχει μη προβλεπόμενος αντίκτυπος. Ε, τα συγκεκριμένα θεσμικά όργανα λοιπόν και ε, ρωτήσατε αν υπάρχει κάποιο κατόφλι ε, σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων. Υπάρχει λόγος που υποβάλλονται αυτές οι δηλώσεις. Να εντοπίζεται και να αποτρέπεται η σύγκρουση συμφερόντων ή να μπορεί να ανοιχνευτεί. Το θέμα λοιπόν ε, σχετικά με τις συγκεκριμένες ε, ε, περιπτώσεις, για παράδειγμα την φιλοξενία, τις προκλήσεις, προσκλήσεις, συγγνώμη, αν, μπορούν, αν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ή όχι. Αυτό θα πρέπει να το δούμε ευρύτερα, διότι πάντα υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο όταν έχουμε μια διοικητική δράση. Θα πρέπει λοιπόν να εξισορροπηθεί η παροχή ε, χρήσιμων πληροφοριών, ε, θα πρέπει να δούμε ε, αυτό σε σχέση με τη σύγκρουση συμφερόντων. Θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι όμως οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του πάνελ. Ινιές, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του πάνελ για την ενημέρωση που μας πρόσφεραν και θα πρέπει και να αναγνωρίσουμε ότι στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που δεν καλύπτονται, δεν είναι ικανοποιημένοι από την ενημέρωση που έγινε. Πάντως εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει οι εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή να έρχονται προετοιμασμένοι και ότι θα πρέπει να περιμένουν ότι θα ανακύψουν τέτοια ζητήματα. Γιατί έχουμε κάποιε συγκεκριμένε περιπτώσει. που έχουν συγκεκριμένα ανακύψει με επιτρόπου και όχι μόνο. Επομένω, θα πρέπει εμπάσχετο οι εκπρόσωποι τη Επιτροπή να έρχονται προετοιμασμένοι για τι ερωτήσει των συνέδρων, του οποίου και ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να κλείσω ευχαριστώντα τον εκπρόσωπο του διότι νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ ας πούμε προέρχομαι από τον Νότο και ε, λένε ότι εκεί ψέματα. Έμαθα όμω ότι τόσο χρόνια που είμαι εδώ ε, βουλευτή. έμαθα πώ λειτουργεί η διοίκηση. Και αντί να ιδιωτικοποιούμε, να εξαθλιώνουμε τη διοίκηση θα πρέπει συνενετικά να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε, να την κάνουμε πιο πιο ισχυρή την ε, διοίκηση. Ούτως ώστε να γεννιούνται ιδέες, προτάσεις. Μην έχουμε μόνο από το εξωτερικό επομένως αυτό το, αυτή την εισφορά ιδεών. και όπως ε, έλεγε ο συνάδελφος από την Βρετανία χρειάζεται μεθοδολογία διάφανη όσον αφορά τις επαφές μας και τη συνεργασία μας με τα λόμπι. Γιατί έχουμε βιομηχανία και έχουμε και την αντιβιομηχανία. Δηλαδή είναι και κάτι άλλο το οποίο έμαθα τώρα και ήταν πάρα πολύ επώδυνο. Αυτό το, το έμαθα αυτά τα χρόνια ότι υπάρχουν εθνικά συμφέροντα και υπάρχουν και ευρωπαϊκά συμφέροντα. Αυτό είναι άλλη προβληματική, άλλου είδους σύγκρουση συμφερόντων. Και μάθαμε επομένως το επώδυνο το ότι θα πρέπει κανείς να δίνει μάχες σκληρές για να εξισορροπήσει τα εθνικά με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα τα οποία είναι περίπλοκα και κάθε φορά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορεί κανείς να κάνει τις διακρίσεις και να καταπολεμεί τους κινδύνους από αυτή την σύγκρουση συμφερόντων. Άρα αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πώς θα προλάβουμε τη σύγκρουση, πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ακαιρεότητα και, να, και την ικανότητα του να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε περίπτωση. Και ο πρόσωπος της Γκρέκο ε, ανέφερε κάποιες χώρες, Πολωνία, Εστονία και εγώ θα μπορούσα να σας δώσω πολλά άλλα παραδείγματα σύγκρουση συμφέροντων με άλλες χώρες ε, και από τα 12 παλαιά κράτη-μέλη, τη Βρετανία, την... Ε, ναι, και, και, το, και το Βέλγιο. Άρα δεν είναι το θέμα η Πολωνία, ε, η Εστονία και η Νορβηγία. Και οι παλιοί έχουμε ε, διάφορα θέματα, διάφορα τέτοια προβλήματα και διάφορα σκάνδαλα. Άλλωστε το σκάνδαλο μπάνκι μορφώσει κάποιον που δεν είναι ούτε στονός ούτε πολωνός. Συνεχώς μαθαίνουμε. Όσο ζούμε μαθαίνουμε και σε ευχαριστώ επομένω και εσάς αγαπητοί ε, μέλη του πάνελ και του συναδέλφου. Παρακαλώ να έρθουν στο ε, Προεδρείο εδώ τα μέλη του δεύτερου πάνελ. Και σα διαβεβαιώ ότι το δεύτερο ήμιση της ακρόασης θα πρέπει να το δούμε σοβαρά. Γιατί όπως είναι τα πράγματα έχουμε μόλις ε, μία ώρα στη θέση μας την και τους διερμήνες. Λείπει κάποιος από το ελεγκτικό συνέδριο. Τι να κάνουμε. Η γρήπη είναι κάτι που τον αντιμετωπίζουμε όλοι. herman jan mee kon Okay, um, Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις ε, προς την ε, Επιτροπή που δεν έχουν ε, απαντηθεί. Θα έλεγα λοιπόν να τις συντάξουμε, να γράψουμε και τη στείλουμε στην Επιτροπή για να μας απαντήσει. Πάμε τώρα στο δεύτερο ε, σκέλος της ακροασής μας. Ο κύριος Χέρμαν που είναι ο συντακτής ε, της απαλλαγής ε, των ε, εξωτερικών οργανισμών. Καλωσορίζω τον κύριο Πολ Ντεκλέρκ από την Alter EU. Κύριε Ντεκλέρκ, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή που μας κάλεσε. Εγώ εργάζομαι για την Friends of the Earth Europe. Είναι περιβαλλοντική οργάνωση στην περίπτωση αυτή βέβαια εκπροσωπώ την Alter EU. Εμείς ε, ασχολούμεθα με θέματα διαφάνειας, ε, σύγκρουσης ε, συμφερόντων που έχουν σχέση με το Κοινοβούλιο, με ομάδες εμπειρογνωμόνων, με επιτρόπους, όλα αυτά κατά τα τελευταία 7,5 χρόνια. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσω να σας πω χρήσιμα πράγματα. Θα μιλήσω για δύο θέματα. Το ένα έχει σχέση με τον χημικό οργανισμό και πώς ακριβώς αντιμετωπίζει τη σύγκρουση συμφερόντων. Και θα ήθελα να ξεκινήσω ε, με κάποια λόγια για το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων στο ίδιο το Κοινοβούλιο κατά το παρελθόν. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα διότι πριν από 1,5 χρόνο ε, θεσπίστηκε ο νέας, ε, νέος κώδικας διοντολογίας για ε, να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με ευρωβουλευτές. Εμείς στηρίζουμε αυτό το νέο κώδικα διοντολογίας γιατί προβλέπει συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να εισαχθούν, να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα Βέβαια, αυτό που βλέπουμε τώρα, 1,5 ε, χρόνο μετά τη θέση σχέφου του κώδικα, βλέπουμε ότι η εφαρμογή του κώδικα δεν είναι δεν υπάρχουν φιλόδοξα σχέδια για να αλλάξει η συμπεριφορά των ευρωβουλευτών. Βλέπουμε ότι ακολουθείται η πεπατημένη και το, το, ο κώδικας αυτός ε, δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωβουλευτές αντιμετωπίζουν ε, ε, ηθικής φύσεως θέματα. Ας δούμε ποια είναι τα βασικά σημεία. Το βασικότερο απ' όλα είναι ότι αρκετοί ευρωβουλευτές δεν παίρνουν στα σοβαρά τον κώδικα αυτό. Εμείς ως φίλοι της γης ε, κάναμε πριν από 6 μήνες ε, μία έρευνα και είδαμε όλες τις 750 δηλώσεις ε, συμφερόντων και διαπιστώσαμε ότι το 12% ήταν κενό, δεν είχαν αναφέρει απολύτως τίποτα. Ένα άλλο 13% των ευρωβουλευτών ανέφεραν ότι πριν γίνουν ευρωβουλευτές ήταν άνεργοι, δεν είχαν επάγγελμα και δεν νομίζουμε ότι αυτό είναι σωστό. Αν λοιπόν προσθέσετε αυτά τα δύο ποσοστά καταλήγουμε στο ότι 25% των ευρωβουλευτών δεν παίρνουν σοβαρά αυτή την υπόθεση του να δηλώσουν τα συμφέροντά τους. Το δεύτερο που διακυβεύεται είναι ότι οι ευρωβουλευτές ε, στην περίπτωση της σύγκρουση συμφερόντων ε, δεν το δηλώνουν αυτό όπως το ζητάει το δικαστήριο. Και ένα 6% των ευρωβουλευτών ε, λένε ότι έχουν μετοχές και συμμετοχές σε ιδιωτικέ εταιρείε. Πάνω από τους μισούς, 55% είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου μιας επιτροπής ε, και πάρα πολλοί βρίσκονται και σε εταιρείε που ε, έχουν συμφέρον σε σχέση με την νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα δηλαδή εδώ υπάρχει το ενδεχόμενο σύγκρουση συμφερόντων. Αν ένας ευρωβουλευτής ε, έχει σχέση με μια εταιρεία η οποία ε, ασκεί πίεση στο Κοινοβούλιο ή αν είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο ή έχει μετοχές μιας εταιρείας που θα επηρεαστεί από την ε, νομοθεσία, είναι σύγκρουση συμφερόντων. Θα αναφέρω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα που υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια και που τίποτα δεν άλλαξε μετά από τον νέο κώδικα δεοντολογίας. Ε, ο κύριος Ρούμπιχ τότε αφού είστε παρόν ακόμα καλύτερα είναι μέλος της ε, Αυστριακής Business Europe αυτός ο οργανισμός ε, κάνει λόμπι. Εδώ λοιπόν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Η περίπτωση αυτή δεν εξετάστηκε από το Κοινοβούλιο. Ένα άλλο παράδειγμα, ο κύριος Λένε, που δεν είναι όμως παρόν, εργάζεται για μια εταιρεία ε, νομικών συμβούλων και αυτή η εταιρεία παρέχει συμβουλές στους πελάτες για θέματα ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτό όμως απαγορεύεται από το νέο κώδικα διοντολογία. Παρ' όλα αυτά δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να πάμε στην προηγούμενη συζήτηση. Χρειαζόμαστε περισσότερους κανόνες ή χρειαζόμαστε εφαρμογή των υφιστάμενων. Νομίζω στις περιπτώσεις αυτές οι κανόνες είναι σαφείς. Το πρόβλημα είναι ότι δεν εφαρμόζονται οι κανόνες. Οι το Προεδρείο του Κοινοβουλίου δεν ε, επιλαμβάνεται αυτών των υποθέσεων. Άλλο παράδειγμα, εμείς ε, καταθέσαμε και πάλι ε, προσφυγή για τον κύριο Ντεχάνε, τον Ευρωβουλευτή, ο οποίος έχει μετοχές στην μεγαλύτερη ζηθοποιία του κόσμου. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ ο κύριος Ντεχάν. Εάν λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λάμβανε αποφάσεις και αυτό ε, θα γίνει στο μέλλον για θέματα όπως είναι η διαφήμιση για εταιρείε συνοπνευματοδών ή η μείωση του ρίου ηλικίας από το οποίο θα μπορούν οι καταναλωτές να αγοράζουν αλκοολούχα ποτά, καταλαβαίνετε αυτό θα επηρεάσει άμεσα την ε, ε, τιμή ε, της μετοχής της ζηθοποιίας αυτής. Πιστεύουμε ότι με το να έχει τόσες πολλές μετοχές ο Ευρωβουλευτής αυτός σε αυτήν την εταιρεία μπορεί να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης, καταγγείλαμε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου είπε και παραθέτω κατά λέξη αυτά που είπε δεν είναι για να παρεμποδίζει τη σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει για να διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα ε, θα πρέπει να δηλώνονται με διαφάνεια. Τέλος παράθεση. Κατ' ουσίαν ο πρόεδρος τι λέει. Λέει ότι ε, αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων πρέπει να αναφέρεται και δεν θα κάνω τίποτα. Δηλαδή ο κώδικας εντολογίας δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο να επιλαμβάνεται αυτών των υποθέσεων. Εφόσον λοιπόν λέμε ότι η εφαρμογή είναι ένα καθοριστικό στοιχείο, απευθύνομαι στο Κοινοβούλιο, δεν ξέρω αν είναι αρμοδιότητά σας, να θίξετε το θέμα με τους αρμόδιους για να κάνουν κάτι. Όχι μόνο να καταρτίζουν ακόμη και με κώδικα και μετά να λένε δεν συμβαίνει τίποτα. Πάμε στην ε, χημική εταιρεία. Πώς αυτή αντιμετωπίζει τη σύγκρουση συμφερόντων. Από το 2011 αυτή η εταιρεία έχει την ε, πολιτική για να αντιμετωπίζει αυτές τις περιπτώσεις και θέλω να σας πω ότι έτσι υπήρξε, υπήρξαν βελτιώσεις. Ε, σαφώς αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και η πολιτική λέει η διαφάνεια είναι το καλύτερο. Επίσης υπάρχει ένας πολύ καλός ορισμός της σύγκρουσης συμφερόντων. Ο ορισμός αυτός λέει όχι μόνο να εξετάζουμε τις περιπτώσεις αλλά και το πώς φαίνονται αυτές προς τα έξω. Επίσης εξετάζονται εξετάζει ενδεχόμενο σύγκρουση συμφερόντων ε, συγγενών. Ε, νομίζω και αυτό είναι καλό. Και βλέπουμε να υπάρχουν όμως και αρκετές ε, ελλείψεις. Πρώτα απ' όλα, το σύστημα σε μεγάλο βαθμό ε, να πόκειται στην ακαιρεότητα ε, του ατόμου, του υπαλλήλου, που καλείται να δηλώσει τα συμφέροντά του ενώ δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος αυτών των δηλώσεων και δεν ε, λαμβάνονται αρκετά μέτρα για να αντιμετωπιστούν τέτοιες ε, περιπτώσεις. Όσον αφορά τώρα την ε, ακεραιότητα των υπαλλήλων. Βεβαίως και μια εταιρεία βασίζεται στο ότι οι υπάλληλοι λένε την αλήθεια. Αλλά δεν αρκεί αυτό γιατί αν ήταν όλοι ακέραιοι, τι να την κάνουμε την πολιτική. Είναι λοιπόν σαφές ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ σε μια έκθεση του 2012 ε, από το ελεγκτικό συνέδριο που έκανε έρευνες αυτό τον, σε αυτή τη χημική εταιρεία και διαπίστωσε ότι ορισμένες ε, δηλώσεις ε, συμφερόντων υπαλλήλων ήταν μέσα σε σφραγισμένους φακέλους που δεν είχαν καν ανοιχθεί. Ε, θα έπρεπε λοιπόν να έχουν εξεταστεί αυτοί οι φάκελοι για να διαπιστωθεί αν υπήρχε ενδεχομένως σύγκρουση συμφερόντων. Δεύτερο πρόβλημα που έχει σχέση με την τρέχουσα πολιτική. Δεν αντιμετωπίζεται σωστά, αντιμετωπίζει σωστά μετακινήσει υπαλλήλων από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα και τα νάπαλιν. Η σύγκρουση συμφερόντων, κατά την άποψή μας, πρέπει να λέει ότι για δύο χρόνια πρέπει να υπάρχει μία πάυση. Κάποιος που εργάζεται για ένα κοινωνικό φορέα δεν μπορεί να εργάζεται για μία ιδιωτική εταιρεία για τα δύο επόμενα χρόνια. Αλλά ισχύει και το αντίστροφο. Έχουμε δει ανθρώπους που έρχονται από τη χημική βιομηχανία και αποκτούν μία θέση σε έναν κοινοτικό οργανισμό. Κατόπιν ε, οι κανόνες για τις μετοχές δεν είναι καλοί. Ο κανόνας λέει τώρα ότι οι υπάλληλοι πρέπει να δηλώσουν αν έχουν μετοχές ε, αξίες πάνω από 10.000 ευρώ σε μία βιομηχανία, σε μία εταιρεία ή τουλάχιστον χημικό βιομηχανία. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί κανείς να σπάσει τις μετοχές του σε διάφορες εταιρείες, και εμείς πιστεύουμε ότι αν ο στόχος είναι να ελέγχονται κάποιοι ε, κλάδοι όπως η χημική βιομηχανία τότε δεν θα πρέπει να υπάρχει καθόλου κανένα συμφέρον σε αυτό τον κλάδο. Άρα δηλαδή θα πρέπει να αναφέρεται ότι κάποιος που κάνει τους ελέγχους δεν θα πρέπει να έχει καθόλου ε, μετοχές ε, σε αυτό τον κλάδο. Υπάρχουν και άλλα θέματα, δεν θα σας τα αναφέρω. Νομίζω ότι αυτή η κριτική που ασκούμε δεν γίνεται μόνο από εμάς. Το ελεγκτικό συνέδριο, σας είπα ήδη, εξέτασε ε, την χημική βιομηχανία αλλά και άλλους φορείς όπως την ΕΦΣΑ και διαπίστωσε ότι όλοι αυτοί δεν χειρίζονται σωστά το θέμα της ε, σύγκρουσης συμφερόντων ο έλεγχος υποψηφίων αναφέρεται ότι οι ε, υποψήφοι υπάλληλοι θα πρέπει να εξετάζονται πριν από την πρόσληψή του, να εξετάζεται επίση μετά την πρόσληψή τους ε, μήπως ήρθανε από τον ιδιωτικό τομέα, ε, να καθοριστεί η ασυμβατότητα. Αυτή είναι η τελευταία πρόταση που θέλω να πω. Απευθύνομαι σε εσά. Αυτές είναι συστάσεις για το ελεγκτικό συνέδριο. Εάν κληθείτε να αποφασίσετε για την απαλλαγή του 2012, παρακαλώ να ελέγξετε εντελεχώς εάν έχουν υπάρξει βελτιώσεις και αν δεν έχουν υπάρξει, σας καλώ και πάλι να μην ε, χορηγήσετε την απαλλαγή του προϋπολογισμού του 2012. Ε, κύριε Ντεκλέρκ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το σίγουρο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ε, φιτιλιάσατε τη συζήτηση. Επόμενος ομιλητής, ε, βεβαίως, αν θέλετε μπορείτε να τοποθετηθείτε σε αυτά που μόλις τώρα ελέγχθησαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά. Ίσως έτσι με καταλαβαίνετε καλύτερα, λέει ο μιλητής. Έχω ετοιμάσει μία ε, παρουσίαση. Ε, θα αναφερθώ έτσι στα θέματα που θέχτηκαν σχετικά με τη δική μας ε, υπηρεσία. Ε, είμαστε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών ε, και έχουμε τέσσερις σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πολίτες. Όπως ε, σας είπα, εφαρμόζουμε τέσσερις ε, σημαντικές νομοθεσίες. Το REACH που υιοθετήθηκε το 2006 μετά από έντονες συζητήσεις εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, έτσι δημιουργηθήκαμε τον Ιούνιο του 2007 και αρχίσαμε να λειτουργούμε κανονικά από τον Ιούνιο του 2008. Όταν μας επισκέφθηκε λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο, ήμασταν ε, τριών ετών, ήμασταν ε, σχετικά νέα ε, υπηρεσία, νέος οργανισμός σε σχέση με άλλους. Επίσης έχουμε την νομοθεσία CLP που υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο το 2008 και εφαρμόστηκε από εμά το 2009 και πέρσι υιοθετήσατε την, εγκρίνατε την νομοθεσία περί βιοκτώνων που μας έδωσε την αρμοδιότητα ε, ε, εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής και πέρσι ε, είχαμε την νομοθεσία περί προηγούμενης ενημέρωσης, το ΠΙΚ. Ποιες είναι οι βασικές μας δραστηριότητες. Ασχολούμαστε με αυτές τις νομοθεσίες ε, διαδίδουμε στο κοινό τις ε, ε, πληροφορίες που συλλέγουμε. Έχουμε δημοσιεύσει περισσότερες πληροφορίες πάνω στα χημικά από οποιονδήποτε άλλο φορέα στον κόσμο. Επίσης, αναπτύσσουμε μόνοι μας τα εργαλεία πληροφορικής που χρησιμοποιούμε και τα διαθέτουμε και σε άλλους που θέλουν να εφαρμόσουν τις ίδιες αρχές. Επίσης, παρέχουμε ρυθμιστική βοήθεια προς την βιομηχανία ε, συντονίζουμε την, εθνική επιβολή, του νόμου σε εθνικό επίπεδο. Πολύ σημαντικό είναι ότι παρέχουμε ε, επιστημονικέ πληροφορίε σχετικά με την χημική ασφάλεια στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό ε, έχουμε το λεπτό θέμα εάν είναι ακέραιες, υψηλής ποιότητας και ανεξάρτητες οι επιστημονικές πληροφορίες. Γι' αυτό από εκεί συνήθως προκύπτει το θέμα της ε, σύγκρουσης συμφερόντων. Εδώ δεν απέχουμε από άλλους οργανισμούς, ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ε, ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας Τροφίμων και εμεί βοηθάμε τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνέ επίπεδο. Τέσσερι στρατηγικού στόχου έχουμε για τα επόμενα χρόνια. Να βελτιστοποιήσουμε την διαθεσιμότητα δεδομένων υψηλή ποιότητα για να επιτρέπουμε την ασφαλή παραγωγή και χρήση των χημικών. Θέλουμε να κινητοποιήσουμε όλες τις ρυθμιστικές αρχές ώστε να χρησιμοποιούν με έξυπνο τρόπο τα δεδομένα αυτά, ώστε να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν είναι τα χημικά που προκαλούν ανησυχίε. Είναι διεθνή υποχρέωση και μέχρι το 2020 ελπίζουμε να έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στο θέμα αυτό. Επίση θέλουμε να αντιμετωπίσουμε επιστημονικέ προκλήσει. επανερχόμαστε εδώ στο θέμα των επιστημονικών συμβουλών και τέλο ε, θέλουμε να ε, ασκούμε πιο αποτελεσματικά τα παλαιά και νέα καθήκοντά μας ώστε να βελτιστοποιήσουμε ε, τη χρήση των πόρων μας ο οργανισμός μας ε, έχει ως εξής ε, και είναι σημαντικό να δείτε ε, το πώς είναι οργανωμένος ο οργανισμός μας. Δεν διορίζουμε μόνοι μας όλα τα μέλη αυτά. Έχουμε λοιπόν το Συμβούλιο Διαχείρισης που διορίζεται από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή την Επιτροπή. Ε, η γραμματεία ε, της οποίας ηγούμε εγώ ε, υπάρχει και εμένα με διορίζει το Διευθυντικό Συμβούλιο. Κατόπιν έχουμε τα, τις επιτροπές στην Επιτροπή των Κρατών Μελών τα μέλη διορίζονται από τα κράτη-μέλη στην Επιτροπή για την αξιολόγηση του κινδύνου και για την κοινωνικο-οικονομική ανάλυση καθώς και στο φόρουμ ε, ε, συγγνώμη, για, τα δύο, για τις επιτροπές ε, τα μέλη διορίζονται από το Διευθυντικό Συμβούλιο ενώ για το Φόρουμ για την Ανταλλαγή Πληροφοριών πάλι τα κράτη-μέλη διορίζουν το, τα μέλη. Πώς μειώνουμε το πρόβλημα της σύγκρουσης συμφερόντων. Σημαντικό είναι ότι προσπαθούμε να είμαστε ανεξάρτητοι και αντικειμενική. Προσπαθούμε δηλαδή κάτι παραπάνω από απλή αποφυγή σύγκρουση συμφερόντων. Ε, ε, διορίζουμε ομάδες, ε, αναθέτουμε σε ομάδες ε, το κάθε θέμα, έτσι δεν υπάρχει ποτέ ένα πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για κάτι. Επίσης έχουμε ευρεία ε, δημόσια διαβούλευση σε κάθε περίπτωση και θα πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη. Κατόπιν ε, υποβάλλουμε τις ε, περιπτώσεις αυτές για γνωμοδότηση ή λήψη αποφάσεων στις επιτροπές μας ε, που θα πρέπει να αποφασίσουν είτε ομόφωνα είτε με μεγάλη πλειοψηφία. Έχουμε, λαμβάνουμε λοιπόν αποφάσεις που βασίζονται στην επιστήμη και που αξιολογούνται από ομότιμους. όσον αφορά την διαφάνεια, ε, ε, τα πρακτικά, αναλυτικά πρακτικά των συνεδριάσεων δημοσιεύονται, ε, εκπροσωπούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς ως παρατηρητές στις επιτροπές και πρέπει να ακολουθούν τον κώδικα θεοντολογίας και επίσης δημοσιεύουν τα, τις μη εμπιστευτικές βερσιών των αποφάσεων διαφάνεια, ευαισθητοποίηση και καλές διαδικασίες είναι λοιπόν σημαντικά για μας. Ε, το θέμα της ε, αποφυγής ε, της σύγκρουσης των συμφερόντων από το 2007 και μετά έχουμε μια πιο απλή πολιτική η οποία υιοθετήθηκε ήδη με την ίδρυση του οργανισμού μας και είχαμε ήδη τότε τους πρώτους κανόνες για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων. Γιατί το είχαμε αυτό ήδη από την αρχή, διότι αυτό το απαιτεί ο κανονισμός ο σχετικός κανονισμός ε, απαιτεί να εργαζόμαστε εμπιστευτικά και ως οργανισμός να έχουμε την εμπιστοσύνη των θεσμικών οργάνων του κοινού ε, και των ενδιαφερομένων. Η νομοθεσία επίσης ε, πιστεύει ότι πρέπει να δημοσιεύονται οι δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων για τα μέλη των Επιτροπών και του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν ε, λοιπόν έγινε αναφορά στα, στις δηλώσεις ε, συμφερόντων ε, των μελών του προσωπικού, είχαμε εμείς κάτι τέτοιο ήδη από την αρχή ως οργανισμός και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, σε κάθε συνάντηση πρέπει σε κάθε συνεδρίαση πρέπει να επαληθεύονται οι ε, δηλώσεις συμφερόντων ε, και συμπεριλαμβάνονται και στα πρακτικά της συνεδρίασης. Έχουμε παρόμοιες ε, ρυθμίσεις για το Συμβούλιο Προσφυγών και έχουμε τους κανόνες αυτούς και για το προσωπικό στο, στο οποίο, στους αναφέρθηκε η Κομισιόν. Επίσης έχουμε κανονισμό σε κάθε έναν από τους φορείς αυτούς, από τις επιτροπές και έχουμε μια νέα πολιτική για τη σύγκρουση συμφερόντων η οποία προχωράει πολύ πιο πέρα από την προηγούμενη διότι ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει σημαντικότερος κίνδυνος έκθεσης ε, της υπηρεσίας μας. Η νέα αυτή πολιτική λοιπόν ε, τι λέει, αναφέρονται οι βασικές αρμοδιότητες και οι διαδικασίες για τον χειρισμό των υποθέσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Επίσης έχουμε και μια συμβουλευτική επιτροπή. Αυτό είναι μοναδικό. Ε, επίσης ε, έχουμε την ειδική ε, έκθεση του ε, Ελεγκτικού Συμβουλίου. Η έκθεση αυτή εκπονήθηκε κατά τη μετάβαση της υπηρεσίας μας από το παλιό στο πιο προχωρημένο σύστημα εξετάσανε λοιπόν το παλιό σύστημα, δεν εξετάσανε το ε, περιεχόμενο και την εφαρμογή του νέου συστήματος, ε, διότι ε, ακόμα το εφαρμόζαμε. Ό,τι λοιπόν και να έχει πει το ελεκτικό συνέδριο για το σύστημά μας, ίσχυε για το παλιό και όχι για το νέο. Γι' αυτό ενημερώσαμε το ελεκτικό συνέδριο ότι έχουμε νέο σύστημα το οποίο είναι πολύ ανεπτυγμένο και έχω υποβάλει και γραπτή έκθεση στο δικό σας πάνελ. Είναι λοιπόν ένα πλήρες νέο σύστημα το οποίο ε, καλύπτει τις συστάσεις ε, του ελεγκτικού συναδρίου και ε, θα ξεκινήσει ο έλεγχος σύμφωνα με αυτό το σύστημα φέτος. Τρεις στοιχές λοιπόν έχει η πολιτική. Πριν, μετά, πριν κατά τη διάρκεια και μετά την ε, ενασχόληση με ένα θέμα. Πριν ε, εξετάζουμε τα ε, θέματα επιλεξιμότητας των μελών. Με άλλα λόγια, δεν βασιζόμαστε μόνο στις δηλώσεις συμφερόντων, υπάρχουν και άλλα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την επιλεξιμότητα των μελών του Διευθυντικού Συμβουλίου και των άλλων επιτροπών, όπου τον διορισμό τον κάνουν άλλοι φορείς, υποβάλλουμε σε αυτούς τους άλλους φορείς ε, τα, τους δικούς μας κανόνες ε, για να μπορούν να τους ε, εφαρμόσουν κατά το διορισμό. Και επίσης έλεγχος το, της σύγκρουσης συμφερόντων συμπεριλαμβάνεται και στη διαδικασία διορισμού νέων προσώπων. Όταν προσλαμβάνουν διευθύνονται συμβούλους θα πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία αυτή. Κατά τη διάρκεια της ε, απασχόλησης, ε, σε αντίθεση με αυτά που υπόθηκαν εδώ, ε, επαληθεύουμε τα, τη δήλωση συμφερόντων με βάση το βιογραφικό των ανθρώπων, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι δηλώσεις συμφερόντων είναι επικαιροποιημένες, επαρκείς και συμμορφώνονται με τα γενικά πρότυπα. Επίσης, ε, εξετάζουμε τις, ε, τη σύγκρουση συμφερόντων ε, σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις και έχουμε και μέτρα διορθωτικά όπου είναι απαραίτητο. Κάθε χρόνο θα πρέπει να ανανεώνονται οι δηλώσεις συμφερόντων, συμπεριλαμβάνουν και τα άλλα μέλη του νοικοκυριού και καλύπτουν την τελευταία πενταετία. Ε, περιλαμβάνουν για παράδειγμα νομική εκπροσώπηση, συμβουλές που δίδονται κλπ. Ε, επίσης ε, σημαντικό είναι το που είναι μέλος κανείς, χρηματοδότηση σε έρευνες κλπ. Άλλα θέματα που αναφέρθηκαν εδώ ήταν η διαδικασία για μετά την απασχόληση. Έχουμε μια αναλυτική τέτοια διαδικασία και για να αναλάβει κανείς σε νέα θέση θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα και ε, εγώ ως διευθυντής μπορώ να, να επιβάλλω περιορισμούς σε περίπτωση που κάποιος θέλει να κάνει αίτηση για δουλειά που συνδέεται με το δικό μας χώρο εργασίας. Ε, στους ε, εξωτερικούς εμπειρογνώμων ε, έχουμε κάποιους περιορισμούς ε, διότι δεν είμαστε εμείς οι εργοδότες τους. Ε, κλείνοντας λοιπόν να πω ότι είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι απέναντι στο θέμα αυτό και ο ε, μπορεί να είναι πολύ σημαντικός. Έχουμε λοιπόν λάβει πολύ πιο αυστηρά μέτρα, εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων όπως και η ΕΜΑ και η ΕΦΣΑ για παράδειγμα νομίζω ότι τα δικά μας πρότυπα είναι κατά 200% πιο υψηλά από αυτά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης εφαρμόζουμε το θέμα της ε, ε, αναλογικότητας ε, και της εφαρμοσιμότητας κατά την κατά τον καθορισμό των διαδικασιών μας έχουμε συμβουλές από, από για να αποφύγουμε ε, ε, συγκρούσεις συμφερόντων. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κατηγορηθεί για πρόβλημα σύγκρουση συμφερόντων. Ελπίζω να παραμείνουν τα πράγματα έτσι. Πάντως, όπως και να έχει, έχουμε συστήματα ώστε να μπορέσουμε να αντιδράσουμε άμεσα σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Και τέλος, ε, το δίκτυο, και, το, το δίκτυο οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ΕΚΑ ε, θα επικροτούσαμε να υπάρχει ε, ευρωπαϊκό σύστημα, να υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα ε, για τις αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, εμείς ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στους πανεπιστημιακούς καθηγητά. εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Μάστερ και θέλω τώρα να μα πείτε κι εσεί τι έχετε να εισφέρετε από τι γνώσει σα για το θέμα. Να σας πω δύο λέξει όσον αφορά το τι έχω πει για, την, ε, για, για το δημόσιο στα κράτη-μέλη, γιατί εγώ έχω εργαστεί ως ε, πανεπιστημιακό σύμβουλος για τι κυβερνήσει επί 7 χρόνια ε, ασχολούμαι με αυτό το θέμα και νομίζω ότι έχω πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα περιοριστώ πάντω το να μην μακρηγορήσω και να μην υπερβάλλω στην παρουσίασή μου. Ε, για να μακρηγορήσουμε. Το πρώτο θα σα ρωτήσω αφορά εσά. Τι νομίζετε. Νομίζετε ότι υπάρχει στον πολιτικό κόσμο, υπάρχει στις ε, δημόσιε υπηρεσίες ή στον ιδιωτικό τομέα Υπάρχει τέτοια ηθική, σαν και αυτή που οποία τώρα συζητούμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να μετρηθεί και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε κατά πόσον υπάρχουν περισσότερε απάντησει, περισσότερα προβλήματα, περισσότερη σεξουαλική παρενόχληση στον ιδιωτικό τομέα όπως στο δημόσιο και σύγκρουση συμφερόντων επίση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι από ό,τι φαίνεται γινόμαστε ε, ολοένα ε, και πιο επικριτική όσον αφορά την ε, συμπεριφορά ε, των, των, των δημοσίων λειτουργών, ολοένα και πιο απαιτητική και λέμε ότι υπάρχουν κάποια τέτοια προβλήματα όσον αφορά την ηθική και ότι τα προβλήματα γίνονται λένε και περισσότερα. Όμως υπάρχουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία έχουμε μια τέτοια κρίση που σοβεί και πρόκειται για, για, για τα ηθικά προβλήματα γενικότερα ε, έχουμε όλο ένα και αυξανόμενο αριθμό περιστατικών. Ε, έχουμε τις πολιτικές ε, που λόγω της κρίσης συρρυκνώνουν. Έχουμε την, τις εταιρικέ σχέσεις δημοσίου δυτικού τομέα. Οπότε έχει γίνει όλο ένα και πιο, και πιο δημοφιλές το να ακολουθεί κανείς τέτοιες στρατηγικές, τέτοιες συνεργασίες. Οπότε και έτσι έχουμε περισσότερες ε, συγκρούσεις συμφερόντων. Όλα ένα και περισσότεροι δέχονται να έχουν μερική απασχόληση ή να δουλεύουν για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο. Και έτσι βλέπετε ότι ε, κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να σκεφτείτε ότι θα πρέπει ε, να, να ρυθμιστεί η σχέση εργασία αυτών των προσώπων, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο αφού θα δουλεύουν μόνο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Άρα έχουμε την ηθική, έχουμε τη συγκρούσει συμφερόντων και διαπιστώνουμε ότι όχι μόνο έχουμε περισσότερες επικρίσεις αλλά και περισσότερες προσδοκίες. Αυτό είναι θετικό. Αλλά εδώ και κάποια χρόνια διαπιστώνουμε ότι έχουμε μια τέτοια έκρηξη ε, των στάνταρ των προτύπων. Περισσότεροι κανόνες, πιο λεπτομερεί κανόνες, πιο πολλοί κώδικες διοντολογίας, πιο ψηλά στάνταρ και όλο ένα και περισσότερα θέματα θεωρείται ότι είναι πια ανήθικα. Περισσότερο από ότι στο παρελθόν το οποίο τα, ξεπερνούσαμε πιο εύκολα. Και γι' αυτό και έχουμε πολύ περισσότερε απαιτήσει όσον αφορά την διαφάνεια. Πιο πολλές επιτροπές αν θέλετε. Οπότε, για τους κανόνες Τι μπορούμε να πούμε. Πρώτα-πρώτα, από ό,τι φαίνεται, κεντρικές και ανατολικέ ευρωπαϊκές χώρες έχουν περισσότερους κανόνες από τις σκανδιναβικές χώρε. Οι σκανδιναβικέ χώρε έχουν τους λιγότερους νόμους και κανόνες. Ε, βλέπετε ότι οι τράπεζες, οι κυβερνητικοί μηχανισμοί ε, έχουν πολύ περισσότερους κανόνες από τα κοινοβούλια. Άρα βλέπουμε ότι κάποιες συγκρούσει συμφερόντων είναι πιο περίπλοκες από άλλες. Έχουμε κάποιες επικουρικές Ε, Ακόμα και τα σχέδια με τα δώρα ε, ρυθμίζονται πάρα πολύ λεπτομέρω. Οπότε τελικά αυτό το οποίο ε, δεν έχει ρυθμιστεί είναι τι γίνεται κατά την περίοδο μετά την απασχόληση. Ε, γιατί να θεωρούμε ότι χρειάζονται περισσότερο κανόνε. Τα περισσότερα κάτι με λένε δεν χρειαζόμαστε περισσότερου κανόνε. Χρειαζόμαστε καλύτερη ε, παρακολούθηση, υποπτία, ε, καλύτερη, καλύτερη διαχείριση και καλύτερη εφαρμογή του νόμου. Αλλά θα, πρέπει να κάνουμε περισσότερα στο, τι, γίνεται, ε, γίνεται με τη σειρώμενη πόρτα, τι γίνεται μετά την απασχόληση τέλο πάντων. Ήδη αυτό δεν συζητήσαμε. Ένα σώρο συγκεκριμένε περιπτώσει. Και είπαμε επομένω τι γίνεται για την αλλαγή δημοσίου με το τομέα. Επομένω αυτό είναι το πραγματικό σημερινό θέμα το οποίο δεν διέπεται από αρκετούς νόμους και κανόνες. Τι θα γίνει με την αποτελεσματικότητα των νόμων. Βέβαια, όσον έχουμε κάποιου άρτιου κανόνε, αυτό δεν έχει να κάνει με το κατά πόσον αυτοί οι άρτιοι κανόνε εφαρμόζονται σωστά. Και επομένω, με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ο κίνδυνο ότι αν έχουμε πολλού κανόνε, ότι και αυτοί οι κανόνε να, να, να, να, να του παραβιάζει κανεί και οπότε χρειάζεται να, να έχουμε πολλού και ενδελεχεί λεπτομέρειε κανόνε και αυτό σε κάποιε χώρε που έχουν ε, πολλού κανόνε, αλλά έχουν υψηλό επίπεδο διαφθορά. και οπότε να πούμε ότι αυτέ οι χώρε που έχουν όλου αυτού του κανόνε, έχουν όλοι, όλα αυτά τα ποσοστά, όλη, όλη αυτή τη διαφθορά αυτό όμω δεν πάει να πει ότι η απορρίθμιση θα είναι μια καλή λύση. τίποτα δεν σημαίνει αυτό. Αυτό που λέμε τώρα σημαίνει ότι, ότι οι κανόνες κάθε αυτοί είναι απλώς ακόμα ένα εργαλείο, σημαντικό εργαλείο, σημαντικό μέσο για την καταπολέμηση των συγκρούσεων συμφερόντων. Και επομένω οι κανόνες από μόνοι του δεν λένε τίποτα. Αυτά. Άλλα δύο πραγματάκια. Τι να πούμε. Ότι υπάρχει ακόμα μια μεγάλη διαφορά μεταξύ Τις θεωρίες και τις πράξεις. Για τα σκάνδαλα λέγονται και γράφονται πολλά, για τη διαφθορά. Πολύ πολύ δραστηριότητα όσον αφορά τη σύγκρουση συμφώνων. Σύμφωνοι, όμως, όμως, όμως, λιγότερα λέγονται και γίνονται όσον αφορά την παρακολούθηση, όσον αφορά Άρα αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να, δούμε πώς θα εφαρμόσουμε αυτά τα οποία προβλέπονται, τα μητρώα, τα πρωτόκολλα, τις επιτροπές. Εγώ μελέτες αξιόλογες δεν έχω ακόμα δει, δεν έχω διαβάσει όσον αφορά την αποτελεσματική λειτουργία των αντιστοίχων ηθικών επιτροπών. Ναι, ναι, για μητρώα υπάρχουν και περισσότερα, όμως, όμως έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αδιαφάνεια όσον αφορά την λειτουργία των διαφόρων επιτροπών. Άρα, εκεί να επικεντρώσουμε ενδιαφέρον μας. Εκεί θα πρέπει να δούμε το, το πώς θα αποκτήσουν θεσμικό χαρακτήρα οι επιταγές της ηθικής. Τώρα, ε, κάτι τελευταίο όσον αφορά ε, τις θεωρίες που κυριαρχούν και την πρακτική. Γι' αυτό που μιλούμε, γι' αυτό που λέμε τώρα, για πολύ κόσμο, είναι μπερδεμένα πράγματα. Σαν την φιλοσοφία του Καντ, ή του Αριστοτέλη. Σημαντικά, αλλά μπερδεμένα. Και αυτοί που είναι στα κέντρα αποφάσεων δεν λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα, διότι δεν μπορούν να, να, να, να συλλάβουν αυτό το περίπλοκο πράγμα που λέγεται ηθική. Αυτό που που χρειάζεται είναι το πώς θα υπάρχει κάποιο είδου δυναμική ε, ηγεσία. Όμως, αν κανείς ρωτήσει τους ηγέτες πώς συμπεριφέρονται στους οργανισμούς, στου φορείς τους, να έχω εδώ πέρα μια παρουσίαση και θα συμπεράνουμε ότι τελικά δεν υπάρχει ηθική ηγεσία. Κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ σοβαρό για φορείς και οργανώσεις. Και θεωρητικά και πρακτικά, επομένως, αυτό ισχύει. Οι ηγέτες να μην διαθέτουν χρόνο για να ασχοληθούν με αυτό το περίπλοκο πράγμα που λέγεται σύγκρουση συμφερόντων. Να, ακόμα και το τι κανόνες, τι κριτήρια χρησιμοποιούν όσον αφορά την πρόσληψη ας πούμε διευθυντών. για τον ορισμό, το διορισμό, την πρόσληψη διευθυντών. Ούτε υπάρχει αντίστοιχη εκπαίδευση, κατάρτιση για το θέμα μας. Υπάρχει εδώ πέρα αυτό το πρακτικό στοιχείο στη σύγκρουση συμφερόντων. Πώς θα αποκτήσει θεσμικό χαρακτήρα αυτή όλη η προβληματική. Δεν, δεν, δεν υπάρχει τέτοια προβληματική. Δεν υπάρχει κάτι ε, το, τέτοιο να έχει θεσμικό χαρακτήρα. Ακριβώς όπως είπε και ο κύριος Τζέικομπ. Άρα το θέμα είναι ακριβώς η υποκτήρια, η παρακολούθηση, η εφαρμογή των κανόνων από την άλλη μεριά. Μαρίτερ, είναι το Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελεύθεσαν ήδη πάρα πολλά ε, και κατόπιν ε, τούτου. Εγώ θα περιοριστώ στο να δώσω ορισμένες πληροφορίες για το τι ακριβώς ε, προτιθέμεθα να κάνουμε στον τομέα των ε, οργανισμών. Εγώ είμαι αρμόδιος για τα θέματα αυτά στην Κομισιόν. Όχι βέβαια απόλυτα αρμόδιος, αλλά διότι κατά κύριο λόγο ασχολούμαι με τους ε, εξωτερικούς οργανισμούς, τα γραφεία. Και όπως θα ξέρετε, πέρυσι μετά από αρκετά χρόνια διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο, Κομισιόν και το Συμβούλιο κατέληξαν σε κοινή ε, προσέγγιση όσον αφορά τους εξωτερικούς οργανισμούς. Σε αυτήν λοιπόν την ε, κοινή προσέγγιση ε, τίθεται το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Κυρίως σύγκρουση συμφερόντων που αφορούν σε μέλη διοικητικών συμβολίων, επιστημονικών επιτροπών, επιτροπών που κατατίθενται προσφυγές και παρεμφερεί. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κοινή προσέγγιση για να προχωρήσει το θέμα αυτό. Και πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Έτσι λοιπόν, με βάση όλα αυτά, η Κομισιόν έλαβε την εντολή να συντάξει χάρτη πορείας για κοινή προσέγγιση. Αυτός ο χάρτης πορείας εγκρίθηκε το Δεκέμβρη του προηγούμενου έτους. Σε αυτό λοιπόν το χάρτη πορείας αναφέρονται πολύ συγκεκριμένες ενέργειες και για φέτο ε, λέμε ότι μία από τις βασικές μας προτεραιότητες είναι να αντιμετωπιστεί το θέμα της ε, σύγκρουσης συμφερόντων. Βεβαίως η ε, πολιτική απέναντι στους εξωτερικούς οργανισμούς. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά κατά κύριο λόγο τους ίδιους τους οργανισμούς, γιατί είναι ανεξάρτητη φορείς. Λέμε λοιπόν στο δικό μας το χάρτη πορείας ότι ε, θεωρούμε ότι όλοι οι οργανισμοί πρέπει κατά τη διάρκεια του έτους να εφαρμόσουν μια σαφή πολιτική σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης ε, να ανταλλάξουν εμπειρίες, να συντονιστούν. Όλα αυτά τα κάνουν ήδη. Οι οργανισμοί έχουν ήδη δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Και επίσης ζητάμε από τους οργανισμούς να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες που ισχύουν για τις επιστημονικές επιτροπές. Αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, το ακούσατε ήδη. Η Επιτροπή λοιπόν δεσμεύτηκε πριν από το τέλος του έτους να καταθέσει ε, κατευθυντήριες γραμμές για τη χάραξη πολιτικής ε, προς αντιμετώπιση περιπτώσεων σύγκρουσης ε, συμφερόντων κυρίως όσον αφορά σε άτομα που εργάζονται σε εξωτερικούς οργανισμούς. Και βεβαίως τώρα βρισκόμαστε μόνο στην αρχή της διαδικασίας. Συζητάμε με τους φορείς, έχουμε συγκεντρώσει τις ε, υπάρχουσες πρακτικές για να υπάρξουμε έτσι, για να αποκτήσουμε μια γενική εικόνα, για να δούμε ε, το τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί έχουν γίνει, να γίνει πάρα πολλά, κυρίως μετά την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχει γίνει πολλή δουλειά σχετικά με τους εξωτερικούς οργανισμούς και θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί τους γιατί επιθυμούμε να καταλήξουμε σε κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν ε, θα είναι εύκολες για τους οργανισμούς και παράλληλα βέβαια θα αποδώσουν και όλα εκείνα τα αποτελέσματα στα οποία προσβλέπουμε όλοι μας. Αν δει την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν ορισμένα βασικά θέματα που πρέπει να ληφθούν ε, σοβαρά υπόψη. Παραδείγματο χάρη, αναφέρεται ότι πρέπει να έχουμε μία προσέγγιση με βάση την ανάλυση κινδύνου όταν καταρτίζουμε πολιτικές για την αντιμετώπιση σύγκρουσης ε, συμφερόντων. Ο κίνδυνος σε σχέση με τους εξωτερικούς οργανισμούς είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το να μιλάμε για έναν εξωτερικό οργανισμό ο οποίος απλά κάνει έρευνα και απλά διαδίδει πληροφορίες. Δεν είναι ίδιες, ίδιοι όλοι οι εξωτερικοί οργανισμοί. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Επίσης, το ελεγκτικό συνέδριο ε, κάνει λόγο για την, τον συστηματικό έλεγχο της σύγκρουσης συμφερόντων και αυτό μέσα από ένα σύστημα δήλωσης των συμφερόντων. Αυτό είναι αξίωμα στο σύστημα. Και η διαφάνεια, κατά την άποψή μας, ε, δεν έρχεται από μόνη της, αλλά είναι ένα καθοριστικό στοιχείο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Επίσης, ε, όπως είδαμε και στη συζήτηση, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ε, δυνατότητες ελέγχου κατά την εφαρμογή των κανόνων. Πρέπει και αυτό να είναι τμήμα των κατευθυντηριών γραμμών. Ε, παράλληλα, ε, πρέπει να καταρτήσουμε κανόνες, οι οποίοι βέβαια να επιτρέπεται να θεσπιστούν, γιατί υπάρχει όλο αυτό το θέμα της μετακίνησης υπαλλήλων από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα και αντίστροφα. Και παρόλα αυτά, οι ε, εξωτερικοί οργανισμοί πρέπει να έχουν πρόσβαση στην βέλτιστη τεχνική γνώση που χρειάζονται. Παράλληλα βέβαια, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι και οι οργανισμοί να είναι σίγουροι ότι δεν αμφιζητούνται οι προθέσεις ή ότι εν πάση περιπτώσει ε, καταβάλλονται προσπάθειες άσκησης επιρροής. Πρέπει λοιπόν και εδώ να εξευρεθεί μια ισορροπία. Προς το παρόν αυτά έχω να σας πω, αυτές είναι οι πρώτες μου απόψεις και μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα δουλέψουμε σκληρά εφέτος για να ε, μπορέσουμε να χαράξουμε μια εφαρμόσιμη πολιτική και να τη δώσουμε αυτή προς εφαρμογή στους ε, εξωτερικούς οργανισμούς. Ευχαριστώ πολύ. Τέσσερις συζήτησαν το λόγο. Μήπως θες να ξεκινήσεις εσύ, Έρμεν. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε μετά την ε, παρουσίαση του κυρίου Ντεκλέρ και σκέφτηκα το, ε, ένα γνωστό λατινικό ρητό που λέει ότι ό,τι επιτρέπεται για το Δία δεν επιτρέπεται για όλους τους ανθρώπους. Είτε μιλάμε για την ε, πολιτική περικαπνού, είτε για την ε, ε σύγκρουση συμφερόντων. Φαίνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακολουθεί αυτό το λατινικό ρητό. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να το σκεφτούμε. Πρέπει να ε, ε, ασκούμε εξίσου πολύ κριτική στους εαυτούς μας όσο και στους ε, υπόλοιπους, όσο και στους άλλους. Δύο ερωτήσεις έχω. Κύριε Ντέμκε, είπατε ότι το πιο, το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι η εφαρμογή, παρακολούθηση και επιβολή των κανόνων. Ποιανού πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η αρμοδιότητα, πρέπει αυτό να γίνει εντός των οργανισμών, θα πρέπει να γίνει εξωτερικά. Και το θέμα των κυρώσεων ε, θύχτηκε από διάφορους συναδέλφους ε, σήμερα. Ε, περιλαμβάνει ε, ακριβώς ε, την παρακολούθηση και την ε, επιβολή του νόμου. Όσον αφορά το ρόλο της ηθικής ηγεσίας, στην πράξη τι ακριβώς σημαίνει αυτό. με παραδείγματα, με αυστηρή παρακολούθηση, με επιβολή πιο αυστηρή εκ των άνω. μπορείτε να μου αναπτύξετε αυτό που έχει να κάνει με τα ηθικά ζητήματα και να μου πείτε εάν εάν είναι κάτι που έχει να κάνει και με τους ίδιους τους κανόνες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να ακολουθήσω και τον ε, προλαλήσαντα. Ε, λείπει ακριβώς αυτή η ηθική ηγεσία, δηλαδή οι άνθρωποι που ε, το προβάλλουν αυτό σε σύνθημα τελικά επηρεάζονται πάρα πολύ από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Νομίζω ότι και ε, συμμερίζομαι τη θέση σας. Ε, έχουμε ε, όμως, ξεφεύγουμε όμως και στη συζήτηση μερικές φορές από τα μέτρα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Ντεκλέρκ. Ε, τα ρίχνουμε όλα στο, στον ίδιο κουβά. Υπάρχει καλό και κακό λόμπι. Θα μου έκανε καλή ε, εντύπωση εάν ε, λαμβάνατε υπόψη τους ε, συναδέλφους που μπορεί να παίρνουν χρήματα από λόμπι και τα λοιπά που δεν συμμετέχουν όμως στις ψηφοφορίες. Και δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο τέλος του δρόμου, δεν έχουμε φτάσει το στόχο μας, αλλά βρισκόμαστε καθοδόν και το γεγονός ότι υπάρχει τώρα πια αυτό ο κώδικας διοντολογία. σίγουρα αποτελεί βελτίωση. Θα ήθελα να πω ότι οι ε, βουλευτές ε, δεν είναι αξιωματούχοι, είναι εκλεγμένοι και οι ε, εκλογείς μου έχουν δικαίωμα να ακουστεί η φωνή τους. Πιστεύω λοιπόν ότι ο κάθε ευρωβουλευτής θα πρέπει να απαντήσει στους εκλογείς τους, στους ψηφοφόρους του αυτό, θέλουν ή όχι. Κύριε καθηγητά και μου έκανε πολύ εντύπωση. Έχετε δίκιο ότι πρέπει να κοιτάξουμε την εφαρμογή. Έχουμε αρκετούς κανόνες. Ε, συμφωνώ με αυτό. Η ερώτηση όμως ε, κατά την εφαρμογή είναι ότι έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Είχαμε την ε, περίπτωση Ντάλι. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε διαφορετικές περιπτώσεις που να τις αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Όσον αφορά την εφαρμογή, δεν νομίζω ότι θα αποφύγουμε τη δημιουργία ενός φορέα. Προς την ΕΧΑ έχω την εξή ερώτηση. Ε, βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Θα ήταν πάρα πολύ καλό εάν τα είχαμε αυτά νωρίτερα. πώς μπορούμε να πετύχουμε τη συμμετοχή των εκπροσώπων του βιομηχανικού τομέα στους οργανισμούς, αλλά με την απαραίτητη διαφάνεια ώστε παντού σε όλους τους οργανισμούς, διότι ε, ε, Πώς μπορούμε λοιπόν ε, να πετύχουμε προς τα έξω να έχουμε τη σωστή εικόνα. Πώς μπορούμε προς τον κύριο Ντεκλέρκ να έχουμε εμπειρογνώμονες από τον βιομηχανικό τομέα, ταυτόχρονα διατηρώντας τα υψηλά πρότυπα που απαιτεί από μας το κοινό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Ντεκλέρκ που ανέφερε το όνομά μου. Πάντα είναι, καλό, πάντα είναι καλή η δημοσιότητα για έναν πολιτικό. Ε, όταν λοιπόν κανείς είναι διαφανής και, διατη... Ε, τηρεί τον ε, κώδικα δεοντολογίας και έχει καλές δηλώσεις συμφερόντων, νομίζω ότι είναι καλό να συζητάμε τι πρέπει να επιτρέπεται για ε, έναν ευρωβουλευτή ή όχι. Εγώ ε, είμαι ε, σιδηρουργό ε, από επάγγελμα, ε, λέμε πάντα ότι πρέπει να χτυπάμε το σίδερο όσο και ακόμα. Ε, είναι, ουσιαστικά εκπροσωπώ τα, συμφέροντα του τομέα μου. Συμμετέχω στο επαγγελματικό επιμελητήριο της Αυστρίας. είναι όλα διαφανή αυτά. Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Σας ευχαριστώ που το αναφέρατε αυτό. Εμένα όμως θα με ενδιέφερε ε, το εξή, διότι είδα το Friends of the Earth ε, ε, ο οργανισμός αυτός έχει 25 ε, ε, ε, εργαζόμενους στις Βρυξέλλες και συμμετέχετε εσείς εκεί. Με τα δικά σας οικονομικά συμφέροντα, τι γίνεται, ποιοι σας χρηματοδοτούν εσάς, δεν βλέπουμε τα νούμερα με την πρώτη ματιά τουλάχιστον και 14 οργανισμούς προωθείται εδώ στις Βρυξέλλες, ε, μεταξύ άλλων ε, μία από τις μεγάλες ενώσεις ε, λομπίστων. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εσείς πώς το χειρίζεστε αυτό εντός του δικού σας οργανισμού και κυρίως για εσάς προσωπικά τις πληροφορίες αυτές που μπορεί να τις βρει κανείς και πώς μπορεί να βελτιώσετε την κατάσταση στο μέλλον. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται για πινκ-πονγκ απλό, είναι ολόκληρο τένις. Κοιτάξτε, βεβαίως και επιτρέπεται κάποιος ε, να εργάζεται σε μια επιχείρηση, να εκπροσωπεί τα συμφέροντά της και είναι και απολύτως ε, θεμητό η εταιρεία αυτή να προσπαθεί να προωθήσει τα συμφέροντά της. Από την άλλη βέβαια η πολιτική έχει και αυτή καθήκον όλο αυτό το θέμα να το χειρίζεται έχοντας κατά νου το κοινό καλό. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν η πολιτική να δέχεται ιδιαίτερα συμφέροντα και να τα προωθεί. Και ακριβώ αυτό τώρα είναι το πρόβλημα και αναφέρομαι λιγάκι σε αυτή την διένεξη μεταξύ κυρίου Ρούμπιχε και Άλτερ. Βεβαίω ε, και πρέπει να ε, αντιμετωπίσει κανεί τον ίδιο τρόπο όλου αυτού του οργανισμού. Μόνο που υπάρχει το ότι το θέμα εδώ εκφράζονται πολύ περισσότερο ιδιαίτερα συμφέροντα από άλλε περιπτώσει. Ε, δηλαδή αν θέλετε εδώ υπάρχει μια σαφή ανισορροπία και ακριβώ αυτή την ανισορροπία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και Έρχομαι τώρα στο ερώτημά μου, που το ερώτημά μου αφορά αφενός την Αλτερ και αφετέρου τον εκπρόσωπο του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, συμφωνώ με αυτά που είπε ο προλαλής σας, δηλαδή πώς ακριβώς ορίζεται η σύγκρουση συμφερόντων. Θα ήθελα να γνωρίζω πώς ακριβώς ε, το ορίζουν αυτό οι εξωτερικοί οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν δείτε λιγάκι τον κώδικα συμπεριφορά, διαπιστώνουμε, αυτή είναι η γνώμη μου, ότι διολυσταίνουμε σε μια νέα σύγκρουση συμφερόντων γιατί δεν είναι δυνατόν, εντάξει αυτό αυτή τη στιγμή δεν αφορά εμά. αλλά α πούμε ε, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου πρέπει να ελέγχει τους ε, συναντέλφου ε, για να διαπιστώσει αν ενδεχομένω κατά το παρελθόν οι ευρωβουλευτέ έχουν υποπέσει σε αυτό το αδίκημα της σύγκρουση συμφερόντων. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ανεξάρτητο οργανισμό για να μπορεί να διαπιστώσει αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων σε ένα θέμα το οποίο είναι είναι και δεν μπορεί να απαντηθεί ξεκάθαρα σε πολλές περιπτώσεις. Και έρχομαι στο τελευταίο μου ερώτημα. Κυρώσεις συγκεκριμένα ε, στον χημικό κλάδο, τι είδου κυρώσει εφαρμόζονται. Και μία άλλη ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της Άλτερ. Οι κυρώσει ε, που προβλέπονται ε, στον κώδικα συμπεριφορά των Ευρωβουλευτών αρκούν ή όχι. Έχουμε ένα δεκαλεπτάκι ακόμα ούτω ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλε τι ερωτήσει. Και οπότε ξεκινούμε τώρα με τον κύριο Ντάνσαρ ε, για τι ε, κυρώσει πέστε μα και επίσης απαντήστε τα σχετικά με, την, το πώ μπορεί να είναι αμερόληπτοι εκπρόσωποι της βιομηχανία κλπ. κλπ. Κύριε Γκρέσλε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Πώς ξεκινάει αυτή η υπόθεση για τη σύγκρουση των συμφερόντων. Συγκρίνουμε τις δηλώσεις με τα βιογραφικά που έχουν υποβληθεί. Και θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη ότι υπάρχει και το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε αυτούς τους κανόνες όσον αφορά την παλήθευση των όσων αναφέρονται στην δήλωση. Όποτε υπάρχει ε, αμφιβολία, έχουμε μια ανεξάρτητη επιτροπή διαβουλευόμαστε με αυτούς τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες που έχουμε όποτε, επαναλαμβάνω, έχουμε ε, αμφιβολίες. Και προβλέπονται κυρώσεις για το προσωπικό. Υπάρχουν πειθαρχικές κυρώσεις σε όλα τα θεσμικά όργανα. Και αυτές οι κυρώσεις επιβάλλονται όποτε συντρέχει κάποια σοβαρή τέτοια περίπτωση συγκρούσεις συμφερόντων. Και αν υπάρχει κάποιο που δεν έχει δηλωθεί, τότε κάποιος αποβάλλεται από τον οργανισμό. Κρίνεται το θέμα από την ε, αρχή, την υπηρεσία, την υπεύθυνη για τον διορισμό και βλέπουμε τι μπορεί να γίνει και κατά πόσον κάποιος δικαιούται να επανατοποθεί τη θέση του εάν υπάρχει κάποιο είδους ε, σοβαρή περίπτωση συγκρόσεως ε, συμφερόντων που δεν έχουν δηλωθεί. Και έτσι αντιμετωπίζεται το πρόβλημα ε, ή πολλές φορές ο προστάμενο ε, συζητεί με αυτόν που έκανε την ε, μη την παράληψη της δηλώσεως και εξασφαλίζεται ότι θα επανελειφθεί το σφάλμα, Εξαρτάται από τη σοβαρότητα και τώρα, όπως σας προείπα, απαιτούμε από αυτού που έχουν υψηλά αξιώματα να δηλώσουν ό,τι συμφέροντα πριν υπογράψουν τη σύμβαση της προσλήψεως. Κατόπιν γίνεται η επαλήθευση και προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο υπάρχουν κάποια, αν πληρούνται τα προϋποθέσεις της ε, επιλεξιμότητας. Εάν έχουμε ε, κάτι το οποίο κατά επανάληψη συντρέχει, τότε δεν προσλαμβάνεται κάποιος. Προσπαθούμε δηλαδή να είμαστε σίγουροι επίσης ότι κάποιο δεν θα κάνει κάποια δουλειά που ισχύει με τη δουλειά που έκανε προηγουμένω. Δηλαδή σε κάποιον άλλο εργοδότη. Και επομένως, εάν κάποιος ε, συνεχίζει και έχει σχέσεις ή έχει ακόμα μια σύμβαση με κάποια βιομηχανία, κάποια επιχείρηση, ενώ δουλεύει για μας, τότε και αυτό αντιμετωπίζεται με τον αντίστοιχο τρόπο. Βεβαίως θα πρέπει όλα αυτά να από αναλογικότητα. Πολύ σημαντικά αυτά και έχουμε νομικούς οι οποίοι έχουν, έχουν εξειδικευτεί στο θέμα μας και οι οποίοι συνομούνται απευθείας με εμένα. Κύριε Δεμκέ, είχατε και από την εισηγήτρια κάποιες ερωτήσεις. Κοιτάξτε, να αρχίσω κάποια διαφορετικά. Όλοι, όλοι έχουμε αλλεργία στη γραφειοκρατία. Όλοι θέλουμε να απαλλαγούμε από τη γραφειοκρατία. Τώρα όμως λέμε για αυτήν την γραφειοκρατία. Άρα θα πρέπει να δούμε ποια είναι η σχέση μεταξύ του να έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία και από την άλλη μεριά να έχουμε περισσότερους κανόνες για να παρακολουθούμε τις σύγκριση Φυσικά και εδώ υπάρχει κάποιο είδου ε, αντίφαση. Το έχουμε ήδη αναλύσει αυτό ε, και έχουμε επίσης μιλήσει και με εκπροσώπους κρατών μελών για το, για το δημόσιο. Τι λέτε, χρειάζεται γραφειοκρατία, ε, επιτροπή διοντολογίας κλπ. Αυτό είναι περίπλοκο, κοστίζει χρήμα χρειάζεται υπαλλήλου κλπ. Από μία διαβούλευση που έγινε, προέκυψε ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω γραφειοκρατία, ότι ελαχίστη, δυνατή. Να μην ε, κάνουμε όπως οι Αμερικανοί. Να μην αποκτήσουμε γραφειοκρατία για τη διοντολογία, για την ηθική. Εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε πολιτικές αποτελεσματικές για τη σύγκρουση συμφερόντων, κάτι χρειάζεται, κάποια γραφειοκρατία χρειάζεται. Ας τη βαφτίσουμε κάπως αλλιώς και θα περάσει. Θα γίνει υποδεκτή. Δεν πειράζει. Δεν είναι τόσο τρομερή αυτή η αντίφαση. Δεν είναι αληθής αντίφαση. Επομένως. Όσον αφορά τώρα τα μητρώα, τα πρωτόκολλα, την εφαρμογή τους, στην Ευρώπη είναι πολύ διαφορετικό το σύστημα. Υπάρχει η προϋπόθεση, η απέτηση για τη δήλωση πολλές φορές είναι άλλοτε είναι τέλο πάντων υποχρεωτικά, άλλοτε όχι, το να, αυτά του είδου τα προαπαιτούμενα, αυτό του είδου υποχρέωση. Στη Σκανδιναβία επίση υπάρχει τέτοια ρύθμιση. Να δούμε τώρα βέβαια πόσο ενδελεχή δήλωση χρειάζεται. Ε, σε άλλε χώρε χρειάζεται πολύ λεπτομερής δήλωση, όπω και στη Ρουμανία, α πούμε, που ζητούν ε, δηλώσει τα πάντα, ακόμα και τι κάνει κανένα με τη γυναίκα του, τι κάνει κανεί στην οικογένειά του, την ιδιωτική ζωή. Υπάρχουν και κάποιο είδου γενικότερε ε, προποθέσει, και μετά το θέμα είναι ποιο διαχειρίζεται, ποιο υποπτεύει τα των αρχείων, μητρών αυτών. αν ρίξετε μια ματιά, στην πρακτική της διοίκησης θα δείτε ότι αυτό είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Αν κανείς να το κάνει στα σοβαρά χρειάζεται κάποιου ειδικού, χρειάζεται κάποιου αφιερωμένους σε αυτό και αυτό λείπει. Δεν έχουμε αρκετούς που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεύτερον, τα περισσότερα θεσμικά όργανα, ιδίω τα κοινοβούλια, έχουν κάποιου αυτορύθμιση, εσωτερικού κανόνε. Η δε εμπειρία έχει καταδείξει μέχρι σήμερα ότι αυτό δεν αποδίδει. Η αυτορύθμιση δεν αποδίδει. Ιδίω τώρα που υπάρχει πίεση από τον κόσμο, από τα ΜΜΕ, Επομένω, ε, μάλλον υπάρχει περισσότερη δυσπιστία παρά περισσότερη ε, αξιοπιστία. Ξέρετε βέβαια για ποιο φορέα, για ποιο θεσμικό όργανο μιλάμε. Πολλέ φορέ. Θα πρέπει να σταθμίσει κανείς και τι πληροφορίε θα δώσει σε κάποιον εξωτερικό πυρογνώμονα. Πάντως, είναι πιο αποτελεσματικό ο εξωτερικός έλεγχο παρά ο εσωτερικός. Και αυτό είναι εμπειρία που προέρχεται από όλα τα μέτωπα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πολ Τεκλέρκ. Ακούσατε διάφορες ε, ερωτήσεις ε, σχετικά με μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, και μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Ακούσατε όμως και ερώτηση από τον κύριο, ένα σμάσο από τον κύριο Ρούμπιχ σχετικά με τους Friends of the Earth, τους φίλους της γης. Στα Ολλανδικά ε, λέμε ότι όποιος ε, πετάει την μπάλα θα πρέπει να την περιμένει, να περιμένει γυρίσει κιόλα. Ε, δεν μου κάνει εντύπωση λοιπόν που απευθυνθήκαν ερωτήσεις προς εμένα. Να ξεκινήσω από την παρατήρηση της κυρίας Κρέσλερ. Είπα ρητά ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων πιθανή σύγκρουση συμφερόντων εάν Ευρωβουλευτή εργάζεται για μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό. Εάν έχετε παραδείγματα λοιπόν ε, παραδείγματα ευρωβουλευτών που ε, εργάζονται παράλληλα για ε, περιβαλλοντικούς οργανισμούς, ναι, πιστεύω ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Το ίδιο βρίσκω να υπάρχει, όπως είπα, στην περίπτωση του κυρίου Ρούμπιχ. Είναι σαφώς ότι ο κύριος ε, Ρούμπιχ ε, και εγώ διαφωνούμε, υπάρχει εδώ διάσταση απόψεων. Εγώ αυτό που έλεγα είναι ότι εργάζεστε για έναν οργανισμό που κάνει lobbying στις Βρυξέλλες για μια σειρά θεμάτων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει καθημερινά αποφάσεις οι οποίες έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για τις οργανώσεις για τις οποίες εργάζεστε. Πιστεύουμε ότι αν είσαστε ε, ευρωβουλευτής με επιρροή και έχετε τέτοια ε, ε, παράλληλη ασχολία, πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνάμει σύγκρουση συμφερόντων. Ε, έχετε επικριθεί ε, για το θέμα αυτό πριν κάποια χρόνια. Δεν είναι λοιπόν καινούριο. Το Κοινοβούλιο ε, έχει υποβάλει νέο κώδικα δεοντολογίας και τίποτα δεν έγινε. Γι' αυτό ακριβώς είναι τόσο σημαντική η επιβολή του νόμου, η εφαρμογή. δεν έχει κανένα νόημα εάν το Κοινοβούλιο θετήσει νέο κώδικα δεοντολογίας χωρίς να το χρησιμοποιήσει. Όσον αφορά την ε, δική μας ε, διαφάνεια, σας καλώ να κοιτάξετε την ιστοσελίδα μας. Ε, μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες. Είμαστε καταχωρημένοι στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Διαφάνειας, όπου δίνουμε πολλές πληροφορίες σχετικά με το πώς ε, ασκούμε πίεση, πώς κάνουμε lobbying, δηλαδή εμείς οι φίλοι της γης. Ε, έχουμε μακρύ κατάλογο των, ε, των δραστηριοτήτων μας, ε, των δαπανών μας ε, για το lobbying. Οι οικονομικοί μας πόροι επίσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα. Θα βρείτε ακριβώς από πού προέρχονται τα χρήματα των φίλων της γης. Εάν είναι δημόσια ή ιδιωτική πηγή, εάν είναι ιδιωτική χορηγία ή αν είναι από τη τις ε, συνεισφορές των μελών μας. Υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές. Ε, θέλατε τις, ε, τη, τα, τα προσωπικά μου οικονομικά συμφέροντα. Ευχαριστώ να σας πω από πού πληρώνομαι. Ωστόσο πιστεύω ότι υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα σε μένα που εργάζομαι για μια οργάνωση λόμπι και εσείς που είσαστε εκλεγμένος αξιωματούχος που υιοθετεί νομοθεσία που αφορά όλους μας. Νομίζω ότι έχετε ευθύνη να δηλώσετε τα οικονομικά συμφέροντα. Δεν λέω ότι δεν το κάνατε, διότι έχουμε δει τη δήλωσή σας, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει διαφορά εδώ. Πιστεύω ότι έχετε ειδική υποχρέωση να, μην, να αποφύγετε την σύγκρουση συμφερόντων στη θέση που κρατάτε όσον αφορά τις ε, κυρώσεις, κύριε Και αρκεί ο κώδικας ε, του Κοινοβουλίου. Δεν ε, πιστεύουμε ότι αρκεί. Όταν γινόταν η συζήτηση για τον κώδικα διοντολογίας, οι κυρώσεις του Ευρωκοινοβουλίου βρέθηκαν να είναι αρκετά αδύναμες. Η μέγιστη ποινή για έναν Ευρωβουλευτή είναι να μην μπορεί να ψηφίσει για δύο εβδομάδες δεν είναι καμιά σοβαρή ποινή αυτό ε, και μετά από αυτό ο Ευρωβουλευτή μπορεί να συνεχίσει να κάνει ό,τι θέλει όπω πριν. Ε, ήταν δύσκολο σε τόσο χρονικό διάστημα να συμφωνήσετε πάνω σε πιο ισχυρέ κυρώσει, αλλά ε, αν αρκετοί ομιλητές, ε, εφόσον αρκετοί ομιλητέ τόνισαν την ανάγκη για πιο αυστηρέ κυρώσει, νομίζω ότι το Κοινοβούλιο καλά θα έκανε να τι κάνει πράγματι πιο αυστηρέ. Δεν νομίζω ότι, έγιναν, ότι απευθύνθηκαν ερωτήσεις απευθείας ε, στον κύριο Τενρέιρο. Ε, ε, να κλείσουμε τώρα, ακούσουμε πρώτα τον Χέρμαν και μετά την Ίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Ώστε να κλείσουμε γρήγορα τη συνεδρίαση, καταρχήν φοβάμαι ότι η πολιτική από μόνη της έχει ένα μόνιμο πρόβλημα σύγκρουσης συμφερόντων, διότι η πολιτική ε, είναι ουσιαστικά επιλογή συμφερόντων και γι' αυτό είναι αιώνιο το πρόβλημα αυτό. Πιστεύω ότι στην πολιτική όσον αφορά την πολιτική συμφερόντων υπάρχει πρόβλημα εάν υπάρχουν προσωπικά συμφέροντα και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Άκουσα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα το πρωί. Είμαι πεπισμένος ότι η εξωτερική παρακολούθηση είναι πάρα πολύ σημαντική στα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς μπορούμε να χειριστούμε το θέμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άκουσα τον εκτελεστικό διευθυντή της ΕΚΑ και αντιλαμβάνομαι ότι η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σε κάποιες περιπτώσεις είναι ήδη ε, ξεπερασμένη. Την έλαβαμε στο τέλος ε, της προηγούμενης χρονιάς, ε, αλλά ήδη το καλοκαίρι υπήρχαν σχέδια του νέου συστήματος. Και έχω ακούσει όχι μόνο από την ΕΚΑ που μας κάνατε την παρουσίαση, αλλά και από άλλους οργανισμούς ότι ε, τα όσα έχουν γίνει μετά τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου. Είναι σημαντικά και ότι η καθυστέρηση της ε, απαλλαγής ε, θα πρέπει να εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από την πρόοδο που έχει σημειωθεί έκτοτε. Οι μεμονωμένοι οργανισμοί λοιπόν μπορεί να προοδεύουν πολύ καλά και τότε δεν βλέπω το λόγο να ε, ε, ε, ε, υπάρξει επιμονή στο θέμα. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Ε, σημείωσα ότι επιτρέπονται παρατηρητές στις επιστημονικές συναντήσεις της ΕΧΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών. Ε, μάλιστα πιστεύω περισσότερο στη διαφάνεια παρά στους νέους κανόνες. Εάν επιτρέψουμε σε όλους ε, να γνωρίζουν τι ακριβώς ε, γίνεται, αυτό μπορεί να επηρεάσει πολύ θετικά όλη τη διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω εδώ. Ίνες, Ίνες έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά εγκριμής. Θα φύγουν στις και 22. Ακούσαμε όλα αυτά και κύριο σας είπα, Θα πρέπει να διαλέξουμε επί τη βάση αυτών των κριτηρίων. Γιατί έχουμε τους ομιλητές από τρεις φορές που ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται με το λόμπι και ακούσαμε και τους φίλους της γης μας τα είπαν επομένως. Και υπάρχει δρόμος αρετής και κακίας και για τα λόμπι. Και όταν τελικά αποφασίζουμε να συρρυκνώσουμε την διοίκηση και στο επίπεδο κράτους και σε επίπεδο Ευρώπης, τότε πώς θα έχουμε τις εγγύσεις που θέλουν οι Ευρωπαίοι. Δεν λέω γραφειοκρατία, λέω η διοίκηση. Η γραφειοκρατία είναι η αρνητική πτυχή. Οπότε τη σήμερα ημέρα με όλη αυτή τη λιτότητα δεν είναι τυχαίο το ότι έχουμε τη συρρήκνωση της διοίκησης οπότε και έτσι ποιος γίνει κερδισμένο, κάτι εξωτερικό στην Ευρώπη η δικηγόροι, τα δικηγορικά γραφεία και σιγά σιγά θα γίνει αυτό και σε εμά στην Ευρώπη. Έχουμε εδώ και τις συγκρούσεις βορρά-νότου, αλλά υπάρχουν επομένως και κάποιες άλλες πτυχές σημαντικές. Χρειάζεται να υπάρχει ο έλεγχος είναι κάτι το υπαρκτό η σύγκρουσεις των σημαντών. Άλλωστε όλοι είμαστε αρκετά όριμοι για να ξέρουμε μέχρι που θα φτάσουμε πέρα από την απλή αντιπαράθεση. Γιατί έχουμε μια θητεία τετραετή και δεν μπορούμε ε, ενδιάμεσα από τη μία θητεία ή την άλλη ενδιάμεσα να αδρανούμε πέρα από τις ε, εξτοτίες που γίνονται από το το ΜΕ, ούτως ώστε να μπορούμε να βρούμε κάποια σωστή λύση. Θα πρέπει να ενεργηθεί η πόρτα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή να υπάρχει διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι κάτι το... αφορά όλο τον κόσμο, είναι κάτι το δημόσιο, ούτως υπήν. Βέβαια, είναι δύσκολη διαχείριση πολλά πράγματα, είναι υπερβολικά τεχνικά, τεχνοκρατικά. Βέβαια από την άλλη μεριά δεν μπορεί κανείς να δουλεύει σαν ήταν μάντης. Πάντως αυτό ισχύει και για τις ε, διάφορες υπηρεσίες που νομίζω ότι έχουν καταβάλει πολύ σημαντική προσπάθεια. Και οι εμπειρογνώμονες έχουν ε, πείρα από την ε, σύγκρουση συμφερόντων και από το πώς μπορεί να ε, υλοποιηθεί η προσπάθεια που γίνεται σχετικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αυτό το φύλλο μας έδειξε κάποιες ε, κατευθύνσεις και έτσι μπορούμε να δούμε ο καθένας τι ευθύνες έχει, ποιες οι υπηρεσίες, ποιες οι κομισιόν. Εμεί πάντοτε θεωρούμε υπεύθυνη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάντοτε ζητούμε να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και με τι ε, περιφερειακέ υπηρεσίε. Επομένω, όσον αφορά του κανόνε και την εφαρμογή του, θέλουμε να υπάρχουν οι κυρώσει και για το δημόσιο και κοινωνικέ ε, κυρώσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά πάντως το σίγουρο ότι χρειάζεται έλεγχος σε κάθε υπηρεσία, σε κάθε διοίκηση να υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί. Όπως σωστά μας τα είπε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, ότι θα χρειάζεται ίσως για περισσότερο έλεγχο, περισσότερο προσωπικό. Γιατί πάντοτε, πολλές φορές, αν ψάξει κανείς, βρίσκει. Και στο, στην αντιπαράθεση των συμφέροντων και μέσα στην, στο πλαίσιο της Ευρώπης. Πολλά συμφέροντα. Αλλά ακριβώ όπως προέκυψε, και έχουμε την έκθεση τη δική μου και του κύριου Γκερβάντη, όπου μπορούμε όλα αυτά τα οποία ακούσαμε και εκτό από τι ερωτήσει και κυρίω τι απαντήσει που ακούσαμε να τι ενσωματώσουμε. Ευχαριστώ για όλα όσα είπατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και αυτό το δεύτερο πάνελ. Νομίζω ότι το δεύτερο τμήμα ήταν ε, πολύ ενδιαφέρον, όπως και το πρώτο. Ευχαριστούμε πολύ τους διερμηνείς. Γεια σας.